may ask you to take seat. Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε με την ακρόασή μας. Θα ήθελα όσοι παρευρίσκεστε να, να κάθεστε στις θέσεις σας, όχι σε θέση άλλων και μπορείτε να παρακολουθήσετε την ακρόαση από την αίθουσα ακρόασης και μέσω της ε, ιστοσελίδες μας και μόνο τα μέλη μπορούν να χειροκροτούν. Καλημέρα σας. Η κυρία Ολσφογκ είναι πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και ο κύριος Μπούζεκ από την Επιτροπή ε, Ενέργειας, Έρευνας και Περιβάλλοντας και εγώ από την Επιτροπή ΕΚΟΝ θα ήθελα να καλωσορίσουμε τον κύριο Κατάινεν ο οποίος ε, είναι υπεύθυνος ή θα είναι υπεύθυνος για την απασχόληση, ανάπτυξη, επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα. Εάν λοιπόν και επειδή το χαρτοφυλάκιο ε, σχετίζεται με την εργασία των ε, επιτροπών αυτών, ε, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η γνώμη τους. Επίσης, ε, εμπλεκόμενες επιτροπές είναι η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και η Επιτροπή Μεταφορών. Συνεπώς, θέλουμε οι επιτροπές να κρίνουν κατά πόσο ο υποψήφιος επίτροπος μπορεί να είναι μέλος του διευθυντηρίου και να αναλάβει το εν λόγω χαρτοφυλάκιο. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι πριν από την ακρόαση ο υποψήφιος επίτροπος απάντησε γραπτό σε ένα ερωτηματολόγιο το ερωτηματολόγιο έχει μεταφραστεί σε όλες τις κοινοτικές ε, ε, γλώσσες και επίσης έχει υποβάλει και μία δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Η Επιτροπή Γιούρη δεν έχει παρατηρήσει ως προς τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων του υποψηφίου επιτρόπου. Ο υποψήφιος επίτροπος θα προβεί σε μία εισήγηση 15 λεπτών και στη συνέχεια θα, έχουμε 5, θα διαθέτει μάλλον 5 λεπτά για μία καταλεκτική δήλωση. Μετά θα υποβληθούν 45 ερωτήσεις από τους ε, Ευρωβουλευτές. Ένα λεπτό η ερώτηση και δύο λεπτά η απάντηση από τον υποψήφιο επίτροπο. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους ευρωβουλευτές ότι η αρχή των τριών λεπτών θα εφαρμοστεί αυστηρά. Υπάρχει διερμηνία σε 23 γλώσσες, άρα όλοι οι ομιλητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη μητρική τους γλώσσα. Και μπορείτε να παρακολουθήσετε την ακρόαση από την ιστοσελίδα μας. Ως πρόεδρος ΣΥΚΟΝ θα ήθελα να κάνω ορισμένα εισαγωγικά σχόλια θα πρέπει η νέα Επιτροπή να φτάσει σε φιλόδοξους στόχους μέσα στα πλαίσια της ανάκαμψης, της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της όθησης της εργασίας στην πραγματική οικονομία. Λαμβάνοντας υπόψη και την κρίση που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια. Άρα το πακέτο των 300 δις που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Γιούγκερ για ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις ε, σχετίζεται με το όλο θέμα και θα ακούσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ε, όπως αναφέρεται στην ε, επιστολή, αφορά την, ε, τις υποδομές, έρευνα, καινοτομία και υποδομές, έτσι ώστε οι άνεργοι να επανέλθουν στην αγορά εργασίας με αξιοπρεπή εργασία. Επίσης, με την εγγύηση για τους νέους θα πρέπει να βοηθήσουμε τους νέους και ε, τη χρησιμοποίηση των δεξιοτήτων τους. Το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συντονίσουν αυτές τις δραστηριότητες λαμβάνοντας υπόψη τη, τον κοινωνικό αντίκτυπο της διαρθρωτικής ε, μεταρρύθμισης μετά την απόφαση των συντονιστών της Επιτροπής ΕΚΟΝ ε, ζήτησα περαιτέρω διασαφήσεις από τον πρόεδρο Γιούγκερ σε σχέση με τον επιμερισμό ευθυνών στον οικονομικό τομέα σε σχέση, και ιδιαίτερα σε σχέση με την εξωτερική και εσωτερική εκπροσώπηση της Επιτροπής και αναμένουμε τις απαντήσεις του ε, Προέδρου. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαρίτα Ούσεμπογκ. Ευχαριστώ, θα μιλήσω στα Σουηδικά. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις στον οικονομικό τομέα. Έχει μεγάλη σημασία να προωθήσουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση για να προωθήσουμε όμως αυτές τις ε, δραστηριότητες, δεν θα πρέπει να υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός και θα πρέπει οι μισθωτοί, οι εργαζόμενοι να την χάνουν προστασίας. Μία πραγματική αγορά δεν θα πρέπει να ε, συρρυκνώνει την αγορά και τις συλλογικέ συμβάσεις. Δεν θα πρέπει να υπάρχει συρρύκνωση ή παλινοδία και ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών ε, μελών, διότι υπ' αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομένων και να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά, να λειτουργήσει σωστά η αγορά εργασίας. Επίσης, οι ιδιαίτερα χαμηλοί μισθοί δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί. Βλέπουμε ότι ανακύπτει εθνικισμός και λαϊκισμός, όλο ένα και περισσότερο. Γι' αυτό κύριε Κατάινεν, είναι πολύ σημαντική η θέση σας και το χαρτοφυλάκιό σας. Άρα η λέξη απασχόληση είναι πολύ σημαντική μέσα στα πλαίσια του χαρτοφυλακίου σας. Ευχαριστούμε την κυρία Μαρίτα ε, Ουλσκοκ και τον κύριο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη. Σας ευχαριστώ που συμπροεδρεύετε σε αυτή την ακρόαση είναι η τελευταία μέρα των ακροάσεων και αυτό είναι ένα καλό νέο για τους ευρωβουλευτές. Παρευρεθήκαμε σε πολλές ακροάσεις. Έγιναν πολλές συζητήσεις για τα ευρωπαϊκά ε, θέματα. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Γιούρκη Κατάινεν που ε, είναι υποψήφιος αντιπρόεδρος για τη νέα Επιτροπή και να καλωσορίσω όλους τους συναδέλφους από την ε, ΕΚΟΝ, την Επιτροπή Απασχόλησης και ε, όλους τους εκπρόσωπους των ΜΚΟ, ΜΜΕ, Βιομηχανίε και κράτη-μέλη. Πρόκειται για μια δημόσια ακρόαση την οποία μπορούν να παρακολουθήσουν οι πάντες. Θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια, γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να μπορείτε να παρακολουθήσετε την ακρόαση στο διαδίκτυο. Θα ήθελα να πω κι εγώ ορισμένα λόγια για τη δική μου επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την έρευνα, καινοτομία ε, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα, ΜΜΕ, ενέργεια, ψηφιακή οικονομία. Όλα αυτά τα, όλες αυτές οι συνιστώσεις ε, προωθούν την ανταγωνιστικότητα και εμπίπτουν στους τομείς ε, του υποψηφίου επιτρόπου, που θα πρέπει να συντονίσει και με άλλους επιτρόπους. Μέσα στα πλαίσια του χαρτοφυλακίου του έχουμε πολλές προκλήσεις για την επόμενη πενταετία σε όλους αυτούς τους τομείς και οι συνάδελφοι από την Ήτρε, την οποία εκπροσωπώ, θέλουν να γνωρίσουν πόσο ο υποψήφιος επίτροπος προτίθεται να ανταποκριθεί δηλαδή να ανταποκριθεί στις ε, προσδοκίες των ε, πολιτών. Θα ήθελα τώρα ο κύριος Γκουαλτιέρη να αναλάβει την ακρόαση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπούζεκ. Ο κύριος Κριστιανής Κάρινς έχει το λόγο. Δεν είναι σκόπιμο να ακούσουμε πρώτα τον Επίτροπο.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 και η ολοκλήρωση οδήγησε σε σταθερότητα. Ως Πρωθυπουργός ήμουνα επικεφαλής έξι ε, κυβερνητικών ε, συμμαχιών, κυβερνήσεων συνασπισμού που συμμετείχαν πράσινοι σοσιαλιστές, ε, η αριστερά, η φιλελεύθερη και το ΕΛΚ. Το να είναι κανείς πρωθυπουργός δεν σημαίνει ότι είναι πραγματικά επικεφαλής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 τα αποτελέσματα. Ως πρώην Πρωθυπουργό μια κυβέρνησης συνασπισμού που απαρτιζόταν από έξι κόμματα, μου είναι γνώριμη αυτή η εργασία. Ένα πολύ καλό παράδειγμα θα είναι το πακέτο επενδύσεων. Θα ήθελα να ε, λάβω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 Thank you, Mr. Commissioner Σε ευχαριστούμε κύριε υποψήφιε επίτροπε. Τώρα ξεκινάμε με τον πρώτο γύρο ομιλητών και ξεκινάμε με τον Χριστιαν Σκάρινς, ε, συντονιστής της Ήτρε από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Κατάινεν. Δουλειές, ανάπτυξη, επένδυση και ανταγωνιστικότητα. Τέσσερις λέξεις που προκαλούν σιελόρια σε όλους τους πολιτικούς. Όλοι υπέρ είμαστε, αλλά βεβαίως το ερώτημα είναι πώς θα επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Αναφέρατε στην εισαγωγή σας ε, και το ανέφερε και ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ένα πακέτο επενδύσεων 300 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα κινητοποιήσει ιδιωτικά και δημόσια κονδύλια. Θα ήθελα λίγο να μπούμε στις λεπτομέρειες. Τι ρόλο νομίζετε πως πρέπει να έχει ο δημόσιος τομέας, τι ρόλο ο ιδιωτικός Και δεύτερον, αυτή τη στιγμή έχουμε αυτά τα κονδύλια που θα πρέπει να επενδυθούν, ποιε πρέπει να είναι οι προτεραιότητε. Μήπως η πρώτη προτεραιότητα θα πρέπει να είναι οι υποδομές για ενέργεια και τηλεπικοινωνίες. Ποιε είναι οι απόψει σας. Ευχαριστώ κύριε Κάριν, στο ερώτημά σας ε, αφορούσε το πού θα βρούμε τα λεφτά και πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Να είμαι σαφής. Ε, χρειάζεται μια νέα όθηση για δουλειές, ανάπτυξη και επενδύσεις. Ε. Δεν είναι μόνο ζήτημα ρευστότητας, αλλά και ζήτημα επενδύσεων. Γιατί αυτό βεβαίως είναι προϋπόθεση για πραγματικές θέσεις εργασίας. Και θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για να μεγιστοποιήσω τον αριθμό θέσεων εργασίας. Γι' αυτό ακριβώς αναφέρατε όντως τους τομείς ε, στους οποίους πρέπει να χρησιμοποιηθούν τηλεπικοινωνίες, μεταφορές ε, και τέτοια πράγματα. Ε, παρά το ότι το μεταξύ κομισιών δεν έχει ακόμα αναλάβει καθήκοντα, εργαζόμαστε με τον πρόεδρο Γιούνκερ για να βρούμε κάποιες επιλογές για να βρεθούν νέα κονδύλια δημόσια για το πακέτο ταυτόχρονα αναγνωρίζοντας πως δεν υπάρχει περιθώριο για ε, νέο χρέος, υψηλότερο χρέος ή ελλείμματα στα κράτη-μέλη. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω ακόμα όλες τις λεπτομέρειες γιατί η Κομισιόν ε, δεν είχε ακόμα περιθώριο να συσκεφθεί και εγώ με τον ε, πρόεδρο Γιούνκερ ακόμα δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε με τους άλλους συναδέλφους. Και χρειαζόμαστε βεβαίως περισσότερο χρόνο και ισχυρή πολιτική συνένεση και βεβαίως κάποια μέσα ε, μπορεί να ε, έχουν κάποιες ευαισθησίες. Οπότε δεν μπορώ να σας αποκαλύψω όλες τις λεπτομέρειες. Αλλά μιλώντας γενικότερα πρέπει να προωθήσουμε και την ζήτηση και την προσφορά. Να μοχλεύσουμε τον προπολογισμό της Ένωσης, να αυξήσουμε τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και να επενδύσουμε στο μέλλον και να έχουμε μια καλύτερη ενιαία αγορά για να αυξηθούν οι ε, ιδιωτικές επενδύσεις. Σας ευχαριστώ. Μαρία Ζωά Ροντρίγκες για τους ε, σοσιαλδημοκράτες. Καλημέρα κύριε Κατάινεν. Χρειαζόμαστε πραγματική αλλαγή στην Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω αν δεσμεύεστε για τα εξή. Πρώτα απ' όλα, η πρώτη προτεραιότητα δεν πρέπει να είναι η γρήγορη εξυγίανση των δημοσιονομικών, αλλά οι επενδύσεις και η δημιουργία θέσεων εργασία. Δεύτερον, αυτό θα απαιτήσει επενδύσεις μεγάλη κλίμακα, όχι μόνο ιδιωτικέ, αλλά και δημόσιε. Τρίτον, χρειάζεται ένα περιθώριο ελιγμών δημοσιονομικών αλλά και ισχυρότερα ευρωπαϊκά μέσα για να στηρίξουμε τις επενδύσεις. Δηλαδή ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Και τέταρτον, οι περισσότερες μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να αφορούν την καινοτομία, την εκπαίδευση για να προσθέσουμε προσθέμενη αξία και να δημιουργήσουμε περισσότερες και καλύτερες δουλειές σε μια πιο έξυπνη, πιο πράσινη κοινωνία. Συμφωνείτε με αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας. Αφορούσε το εάν θα πρέπει να ε, δώσουμε προτεραιότητα στις ε, επενδύσεις αντί στους ισορροπισμένους ε, προϋπολογισμούς για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη. Συμφωνώ με αυτό το οποίο λέτε. Πράγματι ξεπεράσαμε την κατάσταση στην οποία χρειαζόταν να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη ε, στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Δεν είμαστε πια σε συνθήκες πανικού και κατά την άποψή μου περνάμε σε μια νέα φάση αυτή τη στιγμή στην οικονομία για να προσανατολιστούμε προς το μέλλον, να δώσουμε βάρος στις επενδύσεις. Ο Πιέρ είπε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν είχε έρθει εδώ για την ακρόαση, πώς χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις και όσες δημόσιες επενδύσεις απαιτούνται. Και εδώ πέρα συμφωνώ πλήρως. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση για να μειώσουμε τον αντίκτυπο στο χρέος και στο έλλειμμα. Πρέπει επίσης να μοχλεύσουμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό για να μπορέσουμε να αντλήσουμε στο δυνατόν περισσότερα ωφέλη και εδώ πέρα θα συνεργαστώ στενά με την Κρυσταλίνα. Να αυξήσουμε τη δυνατότητα δανεισμού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αλλά και των εθνικών αντιστοίχων τραπεζών. Επίσης, θα ήθελα να ενθαρρύνω τα κράτη-μέλη μαζί με τον πρόεδρο Γιούνκερ, ε, τα κράτη-μέλη ειδικά που έχουν πλέον άσματα να επενδύσουν ε, στο μέλλον. Θα επενδύσουν και στο δικό τους μέλλον, αλλά θα βοηθήσουν και την ευρωπαϊκή οικονομία. Και μετά χρειαζόμαστε κάποια μέτρα στην πλευρά της προσφοράς, ε, όπως η βελτίωση της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς και να εφαρμοστεί η οδηγία των υπηρεσιών. Θα πρέπει να είναι λοιπόν ένα συνολικό πακέτο. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής η κυρία Σουίνμπορν, συντονίστρια του ECR στην Επιτροπή Οικονομικών. Σας ευχαριστώ. Ε, μετά από την ερώτηση του κυρίου Κάρινς για το σχέδιο αυτό των 300 δισεκατομμυρίων ε, ευρώ για επενδύσεις, είναι μάλλον το πιο σημαντικό σας πρόγραμμα. Αλλά έχω κάποιες ανησυχίες πως ε, δεν θα πρέπει να στοχεύουμε τις επενδύσεις που μπορούν να γίνουν από τον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να στοχεύουν ακριβώς τις επενδύσεις εκείνες που δεν μπορούν να προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις. Το πλαίσιο λοιπόν του προηγούμενου πιλωτικού έργου που αφορούσε τα ομόλογα έργου, το Κοινοβούλιο ζήτησε μια μελέτη που θα συγκρίνει το κόστος χρηματοδότησης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για να μην ανταγωνιζόμαστε αθέμητα τον ιδιωτικό τομέα. Μπορείτε να μας πείτε αν έχετε κάποιο σχέδιο σχετικά ιδιωτικός ε, σε σχέση με τον δημόσιο τομέα. Αν θα δεσμευτείτε στη μόχλευση από τον ιδιωτικό τομέα όπου αυτό είναι δυνατόν. Και επίσης όσον αφορά τον αποτέλεσμα πέρα από τον αριθμό θέσεων εργασίας, μήπως να αξιολογήσετε και το κόστος κεφαλαίου των επενδύσεων αυτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σουίνμπορν. Συμφωνώ πλήρως με αυτό το οποίο λέτε για το ότι οι δημόσιες επενδύσεις δεν θα πρέπει να διώχνουν τις ιδιωτικές. Γιατί και αυτός είναι ο κύριος στόχος μας. Δεν έχει νόημα να χρησιμοποιούμε τα λεφτά των φορολογουμένων ε, ε, για σκοπούς που ε, μπορεί να επιτευχθούν αλλιώ. Και πράγματι εκτιμώ τη δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προηγούμενη θητεία του που προσπάθησε να διασφαλίσει πως ε, όλα τα δημόσια κονδύλια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως καταλήτης για ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτό ζητάμε και εμείς. Γιατί πράγματι ε, η έλλειψη είναι στα δημόσια κονδύλια. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε έξυπνα, παραδείγματο χάρη, τον ευρωπαϊκό προπολογισμό για να μοχλεύσουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια για να εισρεύσουν και περισσότερα ε, ιδιωτικά μαζί με τα δημόσια. Καμιά φορά οι αγορές είναι δειλές όταν μιλάμε για έργα τα οποία είναι πολύπλοκα και μακροπρόθεσμα. Γι' αυτό ακριβώς θεωρώ πως χρειάζονται δημόσια κονδύλια. Γιατί ο ιδιωτικό τομέα δεν είναι έτοιμο να αναλάβει όλου του κινδύνου σε μεγάλα έργα. Και είμαι σίγουρο πω και γνωρίζω πως ε, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπάρχει τεχνογνωσία για το πού είναι το όριο και το πώς ε, ακριβώς ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον συνδυασμό αυτών δανεισμού ε, πιο αποτελεσματικά. Γι' αυτό ακριβώς αναμένω και τη συνεργασία μαζί σας γιατί έχετε εμπειρία σε αυτά τα ζητήματα. να βρείτε τον καλύτερο τρόπο για να χρησιμοποιήσουμε τα δημόσια κονδύλια για να προσελκύσουμε ακριβώς και ιδιωτικά. Σας ευχαριστώ. Ραμόν Τρεμόζα ή Μπαλσές για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Κατάινεν στο Κοινοβούλιο, στις γραπτές σας απαντήσεις δίνεται μέγα βάρος στο μέλλον του επενδυτικού πακέτου και πολλοί από εμά συμφωνούμε μαζί σας. Ωστόσο, οι επενδύσεις προς χάρη επενδύσεων είναι λάθος. Έχουμε παραδείγματα στην Ένωση για αεροδρόμια χωρίς ε, ε, πλάνα, για δρόμους ε, χωρίς αυτοκίνητα και για γέφυρες στη μέση του πουθενά. Ε, τέτοια πράγματα συνεχίζονται δυστυχώς. Πώς θα εξασφαλίσετε κύριε Κατάινεν ότι τα προγράμματα που θα επιλέξετε στο μελλοντικό επενδυτικό πακέτο θα έχουν ευρωπαϊκό ενδιαφέρον όσο αφορά την αξία τους για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη. Και παρακαλώ να μας δώσετε πιο συγκεκριμένα απαντήσεις, γιατί αν θέλετε να σας υποστηρίξουμε θα πρέπει μαζί μας να μοιραστείτε πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τρεμόζα. Η ερώτησή σας αφορά πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το δημόσιο χρήμα πιο αποτελεσματικά, πιο αποδοτικά, να μην δαπανώνται δημόσια χρήματα σε σχέδια τα οποία δεν βοηθούν πραγματικά κανέναν. Εγώ πάντοτε θέλω να μιλάω για χρήματα των φορολογούμενων, γιατί Καμιά φορά μπορεί κανείς να πιστεύει πως τα ευρωπαϊκά χρήματα είναι χρήματα που βγαίνουν από καμιά μαύρη τρύπα. Όμως ε, στην ουσία βγαίνουν από τις τσέπες των ε, συμπολιτών μας. Γι' αυτό και πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική η χρήση τους. Κάθε φορά που βγαίνουμε στο εξωτερικό και βλέπουμε ένα το αεροδρόμιο ή έναν αυτοκινητόδρομο που ξέρουμε πως εν μέρει χρηματοδοτήθηκε από τα χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών, μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Πιστεύω λοιπόν ότι η Κομισιόν εν γέννη έμαθε και από το παρελθόν ότι υπάρχουν καλά παραδείγματα χρήσης ε, του δημόσιου χρήματος. Γι' αυτό και χρειάζεται πάντοτε να γίνεται μια σωστή ανάλυση αντικτύπου ε, και σκοπιμότητας πριν να ξεκινούν μεγάλα προγράμματα. Και αυτό όχι μόνο... Μάλλον και αυτό το οφείλουμε ε, στους φορολογούμενους. Επίσης πρέπει να επιλέξουμε πολύ προσεκτικά τα προγράμματα και τα σχέδια που θα χρηματοδοτήσουμε, αλλά και να κάνουμε κλίση στους, στα κράτη-μέλη ώστε να αποδώσουν και να έχουμε έτσι την, ε, δημόσια στήριξη. Τα προγράμματα λοιπόν θα πρέπει να είναι πολύ καλά προγραμματισμένα από την αρχή, να μπορέσουμε να αποφύγουμε λάθη του παρελθόντος. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, Δημήτρης Παπαδημούλης από την GUNGL. Κύριε Κατάινεν, καλημέρα από την ομάδα της Αριστεράς και από την Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε κάποια μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης παρά τη διαφωνία της Bundesbank. Εσείς συμφωνείτε με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κύριος Ντράγκη ή με, την Bundesbank. Ο κύριος Γιούνκερ προτείνει 100 δισεκατομμύρια ευρώ που λιμνάζουν σήμερα στον ESM να διατεθούν για την ενίσχυση της οικονομίας. Ο κύριος Σόιμπλε έσπευσε να διαφωνήσει με άρθρο στο Σπίγκελ. Τι πιστεύετε εσείς, συμφωνείτε με την πρόταση του Προέδρου Γιούνκερ, ναι ή όχι. Το 2012 ως Πρωθυπουργό της Φιλανδίας πήρατε το βραβείο απουσίας κοινοτικής αλληλεγγύης γιατί μόνο εσείς από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητήσατε και πήρατε πρόσθετη εγγύηση από την Ελλάδα 900 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο εσείς είχατε δίκιο και όλοι οι άλλοι είχαν άδικο και με την ίδια κοινοτική αλληλεγγύη σε εισαγωγικά και νεοφιλελεύθερη σκληρότητα θα πολιτευτείτε και ως αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Thank you very much, Mr. Σας ευχαριστώ κύριε Παπαδημούλη. Δεν θα σχολιάσω την πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αν και θα το ήθελα. Ας πούμε απλά ότι είμαι ικανοποιημένος από αυτό το οποίο έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρέπει να διασφαλίσουμε πως η Ευρώπη θα είναι αξιόπιστη. Ακόμα και μετά από την αξιολόγηση και τα stress test που θα γίνουν ε, για τις τράπεζες. Χρειάζεται λοιπόν ένα τείχος προστασίας ακριβώς για να δείξουμε στον έξω κόσμο πως η Ευρώπη είναι ικανή να υπερασπίσει, να αντιμετωπίσει, με συγχωρείτε, ε, τυχόν ε, αναπάντεχες χρεοκοπίες τραπεζών ή αποτυχίες κάποιων τραπεζών. Ας ελπίσουμε πως δεν θα χρειαστεί κρατική στήριξη από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για τις τράπεζες ή για κράτη-μέλη. Επίσης αναφέρατε το ζήτημα των εγγύσεων. Να σας πω τι συνέβη. Ήμουν υπουργό Οικονομικών το 2011 και είχαμε δεχτεί, η, η χώρα μου με συμμετείχε στα πακέτα βοήθειας της Ελλάδας και της ε, Ιρλανδίας. Εγώ ήμουν υπέρ ε, επίσης ε, και του πακέτου βοήθειας της Πορτογαλίας. Είχαμε εκλογές και κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, οι σοσιαλδημοκράτες παραδείγματος χάρη, υποσχέθηκαν στους ψηφοφόρους πως αν γίνουν κυβέρνηση θα ζητήσουν εγγύησεις. Αυτό είναι γεγονός μετά τις εκλογές ε, συμβιβαστήκαμε. Δεν ζητήσαμε εγγύησεις από την Πορτογαλία, γιατί ε, ε, έτσι ήταν η κατάσταση και μετά είπαμε πως εάν ξαναχρησιμοποιηθεί το EFSF η ε, κυβέρνηση θα χρησιμοποιούσε κάποιες εγγύησεις. Θεωρούσαμε πως δεν θα ξαναχρησιμοποιηθεί το EFSF γιατί ακολουθούσε το το ESM, αλλά παρόλα αυτά προτιμήσαμε να ζητήσουμε εγγύησεις. Σας ευχαριστώ, Reinhard Bütikofer, από την Ήτρε. Καλημέρα σας κύριε υποψήφιε Αντιπρόεδρε. Όσον αφορά το ευρωπαϊκό σχέδιο επενδύσεων, θέλω να ρωτήσω το εξής. Κατάλαβα καλά θα σταματήσει αυτή η λανθασμένη κυριαρχία της λιτότητας στην Ευρώπη και από ποιες πηγές θα πρέπει να προέλθουν τα νέα δημόσια κονδύλια ή δεν θα έχουμε νέα δημόσια κονδύλια. Πόσες επιπρόσθετες επενδύσεις από το δημόσιο τομέα θεωρείται αναγκαίες και τι ρόλο θα παίξουν οι τεχνολογίες αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας για μια μετάβαση χαμηλού άνθρακα και πράσινης ανάπτυξης στο πλαίσιο του επενδυτικού αυτού σχεδίου. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Μπιουτικόφερ. Το ερώτημά σας ήταν από πού θα βρεθούν τα νέα αυτά δημόσια κονδύλια, πόσα χρειαζόμαστε και τι ρόλο θα παίξουν οι νέες αυτές πράσινες τεχνολογίες στη δημιουργία θέσεων εργασία. Πρώτα απ' όλα να είμαι σαφής τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη έχουν ανακτήσει την εμπιστοσύνη που είχαν και πολλές από τις ε, χώρες που ήταν σε επικίνδυνη θέση πριν από λίγα χρόνια έχουν επανέλθει αυτή τη στιγμή στις αγορές. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να είμαι σίγουρος πως η Ευρώπη θα ε, αντιμετωπίσει στεναρά αυτές τις οικονομικές πολιτικές και να μην βρεθούμε στη θέση στην οποία ενα ένα, δύο, τρία, κράτη-μέλη θα προκαλέσουν προβλήματα στα υπόλοιπα. Οπότε πρέπει να συνεχίσουμε με υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική. Ταυτόχρονα όμως χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους για επενδύσεις. Φαντάζομαι πως ε, πολλές από αυτές τα επόμενα 5 με 10 χρόνια θα προέρθουν από τον ιδιωτικό τομέα. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να προσθεθούν σε αυτά και οι δημόσιες επενδύσεις και θα πρέπει ακριβώς να συντονίσουμε την ευρωπαϊκή δράση για να μειώσουμε το ευρωπαϊκό χρέος και έλλειμμα και επίσης να έχουμε κάποιες ε, και από τις χώρες που έχουν ε, πλεονάσματα τρεχουσών συναλλαγών και οι χώρες που δεν είναι σε πλεονασματική θέση πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις δημόσιες δαπάνες για να επενδύσουν στην έρευνα και την ανάπτυξη που είναι προϋπόθεση ε, για να δημιουργηθούν ε, παραδείγματος χάρη νέες πράσινες τεχνολογίες. Επίσης χρειάζεται μια καλύτερη ενιαία αγορά για να ενθαρρύνουμε τις πράσινες τεχνολογίες να μπουν στην αγορά και να αντικαταστήσουν τις παλιές και ερυπένουσες. Σας ευχαριστώ. Ο μιλητής μας ήταν από τους Πράσινους, ο επόμενος είναι ο Στίβεν Γουλφ από το EFTD. Γεια σας, είμαι ο κύριος Οφλίν. Δεν ξέρω αν ο Στίβεν Γουλφ είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Εδώ βρίσκομαι, κύριε Κατάινεν. Λέτε στις γραπτές σας απαντήσεις ότι χρειαζόμαστε πιο ανοιχτή καθολική αγορά εργασίας που να ανταποκρίνεται στη ζήτηση. Εννοείται μέσα στα κρατη και μεταξύ των κρατών μελών και πώς αυτό συνδυάζεται με το όσα είπε ο κ. Κάμερον για κάποιο είδους περιορισμού στην ελεύθερη κυκλοφορία για να συνεχίσει να στηρίζει ως προϋπόθεση για να συνεχίσει να στηρίζει τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βούλφα. Νομίζω πως η ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων είναι βασική αξία της Ένωσης. Είναι μία από τις ιδρυτικές αξίες της Ένωσης. Οπότε θέλω να την υπερασπιστώ την αξία αυτή. Επίσης συμφωνώ με τα όσα είπε ο πρόεδρος Γιούγκερ αλλά και η Μαριάν Τάισεν ε, πέρα της ελεύθερης κυκλοφορίας. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτό ε, ότι όλα αυτά δεν θα βοηθήσουν την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των ανθρώπων. Ε, ξέρω ότι γίνονται κάποιες προετοιμασίες ε, σε επίπεδο ομάδας εργασίας, όπου προσπαθούμε να δούμε, να συζητήσουμε ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα του κάθε κράτους μέλους ως προς αυτό. Διότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να χάσουμε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας ε, ε, χωρίς να δηλαδή υπερασπιστούμε τις βασικές μας αξίες όπως είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων. Αν υπάρχουν κάποια στοιχεία κατάχρησης απλά θα πρέπει να τα διορθώσουμε. Και θεωρώ ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι ένας καλός εταίρος που θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις βασικές αξίες και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Μπάρμπαρα Κάπελ από τους μη γεγραμμένους. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κατάινεν, τα τελευταία χρόνια έδειξαν πως χώρες με υψηλό ποσοστό βιομηχανίας στο ΑΕΠ ε, αντιμετώπισαν καλύτερα την κρίση από άλλες. Παρόλα αυτά χάθηκαν εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η Κομισιόν από το 2012 έχει θέσει ως στόχο να αυξηθεί το ποσοστό ε, της βιομηχανίας στο ΑΕΠ μέχρι το 2020 στο 20%. Η τάση αυτή τη στιγμή όμως είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Το ποσοστό του ΑΕΠ τον Ιούνιο του 2013 ε, μειώθηκε και έφτασε στο 16%. Βλέπουμε πως βιομηχανίες φεύγουν από την ε, Ευρώπη, αλλά βλέπετε ας πούμε ότι η First Alpine στην Αυστρία έστειλε μέρος ε, της παραγωγής της της ε, ΗΠΑ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει λάβει κάποιες σχετικές αποφάσεις για αυτούς τους στόχους. Θα ήθελα λοιπόν να σα ρωτήσω το εξή: Πόσο ψηλά θα είναι ε, το ποσοστό το οποίο θέτετε εσείς ως στόχο για την επαναβιομηχάνηση της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά αυτό το οποίο λέτε. Εμένα η χώρα μου πάντα έκανε εξαγωγές. Η κοινωνία, η ευημερία της ε, κοινωνίας βασίζεται ακριβώς στα έσοδα που εξασφαλίζουμε από το εξωτερικό εμπόριο. Γι' αυτό ακριβώς ε, και η ανταγωνιστικότητα είναι ο καλύτερος φίλος του κράτους πρόνοιας. Όταν λοιπόν ε, έχουμε μια χώρα στην οποία ε, ο ρόλος του δημοσίου είναι 55% του ΑΕΠ, δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να έχουμε έναν επιτυχημένο εξαγωγικό τομέα. Ξέρω λοιπόν πολύ καλά τι εννοείται και ο πρόεδρος ε, Γιούνκερ το είπε ότι είναι αφελές να πιστεύουμε ότι θα προχωρήσουμε μόνο με νέες ε, υπηρεσίες Βεβαίως τίθεται το ζήτημα του τι είναι πλέον βιομηχανία και τι ε, υπηρεσίες. Υπάρχουν ακόμα παραδοσιακές βιομηχανίες, αλλά περισσότερες εταιρείε τρέφονται προς τη βιομηχανία. Θα ήθελα λοιπόν εγώ να δώσουμε βάρος στην έρευνα και την ανάπτυξη, γιατί είναι ένας από τους τρόπους για να δημιουργήσουμε νέες ε, βιομηχανίες και οι παραδοσιακές βιομηχανίες πρέπει να ανανεωθούν. Επίσης πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη ενιαία αγορά για τις ανανεώσιμες ε, ενέργειες παραδείγματος χάρη. Χρειάζεται επίσης συμφωνίες ελευθεριομπορίου εμπορίου με τις άλλες περιοχές του κόσμου. Επίσης σύνοχη, κοινωνική συνοχή, γιατί δεν μπορούμε να χάσουμε κανέναν άνθρωπο, γιατί χρειαζόμαστε υψηλά εξειδικευμένη εργασία. Οπότε η ανταγωνιστικότητα είναι πολύ μεγάλο ζήτημα και μπορούμε να κάνουμε πράγματα και στο ευρωπαϊκό και στο εθνικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Παύλος από Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε υποψήφιε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ για την εισήγησή σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σε σχέση με το θέμα του συντονισμού πιστεύω ότι ε, υπάρχει ένα πρόβλημα διότι υπάρχει πιστοτική ανεπάρκεια στα κράτη-μέλη κάτι το οποίο θα μπορούσε να επιληθεί με το Capital Market Union, για το οποίο είναι υπεύθυνο ο κύριος Χιλ, ή ε, από τη συμμετοχή των κρατών μελών, κάτι το οποίο ε, αφορά το χαρτοφυλάκιο του κυρίου Μοσχοβησή. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε αυτή την πτυχή της ανάπτυξης. Επίσης, μπορείτε να μας πείτε ποια μέτρα προτείνετε για την όθηση της ανταγωνιστικότητας. Γιατί ένα από τα βασικά μας θέματα είναι ότι πρέπει να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Η ερώτησή σας σχετίζεται με τον συντονισμό με τους άλλους ε, επιτρόπους για να βελτιώσω την ανταγωνιστικότητα και την δημιουργία θέσεων εργασίας και πόσο μπορούμε να προωθήσουμε την ανταγωνιστικότητα. Χρειάζονται επενδύσεις στην εκπαίδευση και την έρευνα. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει σωστή φορολόγηση. Εμείς στη χώρα μου, στα πλαίσια αυτής της κυβερνητικής ε, συμμαχίας, προσπαθούμε να μειώσουμε τη φορολόγηση ε, κατά 6% αλλά αυξάνουμε τη φορολόγηση των μερισμάτων Δηλαδή, αν βγάλετε τα χρήματα από την επιχείρηση, φορολογούνται ή με υψηλή φορολόγηση. Αν παραμείνουν όμως στην επιχείρηση, φορολογούνται πολύ λιγότερο. Και αυτό είναι ένα επενδυτικό κίνητρο. Αυτό προωθήσαμε στη συμμαχική κυβέρνηση, στην κυβέρνηση συνασπισμού με όλα τα κόμματα, όπως σας είπα, από τη δεξιά μέχρι την ε, αριστερά. Τώρα ως προς την ανταγωνιστικότητα τι θα πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε αν διοριστούμε. Θα ορίσουμε καταρχήν τα προγράμματα υποδομών και τι πρέπει να γίνει στην ε, χρηματοοικονομική αγορά και το θέμα της ε, μόχλευσης στην ΕΚΤ. Θα ζητήσουμε λοιπόν από τους άλλους επιτρόπους να ε, συναντηθούμε και να προβούμε σε κατανομή ευθυνών. Άρα δεν θα γίνει όπως πριν, δηλαδή κάποιος προτείνει κάτι και μετά το υποβάλλει στο διευθυντήριο. Αυτό θα γίνεται, ο προγραμματισμός θα γίνεται εξ αρχής και από κοινού. Το πακέτο δεν είναι έτοιμο γιατί δεν συζητήσαμε όλες τις ε, λεπτομέρειες αλλά δεν θα χρειαστεί πολύς χρόνος. Η Ελίζα Φερέιρα από τους ε, σοσιαλιστές. Κύριε Κατάινεν, η δράση σας είναι πιο σημαντική από τα λόγια, γιατί ως Πρωθυπουργό και υπουργό Οικονομικών της Φιλανδίας ήσασταν υπέρ της λιτότητας. Ε, είπατε ότι αυτοί που έσφαλαν θα έπρεπε να το πληρώσουν και ζητήσατε εγγυήσεις από όλα τα κράτη-μέλη, ακόμα και από την Ισπανία, η Ελλάδα χρειάστηκε να δανειστεί για να ανταποκριθεί στη λιτότητα, κάτι το οποίο ζήσαμε και στην Πορτογαλία. Εσείς μιλήσατε για, το, για την ε, ε για την ε, διεύρυνση, με συγχωρείτε, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και είπατε ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για επενδύσεις. Εσείς μιλάτε σήμερα για ε, μία όθηση επενδύσεις. Γιατί το κάνετε αυτό τώρα, από πού θα προέλθουν τα χρήματα. Σας ευχαριστώ, κυρία Φερέιρα. Θα πρέπει να μειώσουμε το χρέος για να φτάσουμε σε ανάπτυξη και πρέπει να προωθήσουμε την ανάπτυξη για να μειώσουμε το χρέος. Αυτό είπε ο Πιέρ Κοβισή την ε, προηγούμενη εβδομάδα και αυτό υπερασπίζομαι κι εγώ. Γνωρίζω ότι έγιναν πολλές θυσίες από τους πολίτες τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα σε ορισμένες κυβερνήσεις και χώρες και ήταν δύσκολο για κυβερνήσεις να προασπίσουν την ε, αξιοπιστία τους. Έπρεπε να δώσουν μεγάλη μάχη για να επανέλθει η εμπιστοσύνη των πολιτών. Αυτό αποτελεί πρόκριμα για να δημιουργηθούν ε, θέσεις εργασίας και να υπάρξει προσέλκυση επενδύσεων. Τώρα έχουμε ανακτήσει αυτή την εμπιστοσύνη και τώρα θα πρέπει να δώσουμε μία μάχη για το μέλλον. Να κάνουμε μία επέλαση στο μέλλον, όπως λέω και εγώ δηλαδή, να προωθήσουμε τις επενδύσεις για τους πολίτες μας. Και η Ευρώπη θα πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστική. Σε, με μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να μπορέσουν να πωλήσουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Δεν πρόκειται για μαύρο άσπρο, δηλαδή αν χρειαζόμαστε δημοσιονομική πολιτική ή ανάπτυξη. Θα πρέπει να ισχύσουν και τα δύο και θα ήθελα να επιλέξω θέματα που μας ενώνουν, όχι που μας χωρίζουν, διότι όλοι αναμένουν μία πολύ καλή συνεργασία από όλα τα πολιτικά κόμματα για να βρούμε τις ε, καλύτερες λύσεις και τα καλύτερα μέτρα για να προωθήσουμε τις επενδύσεις. Η Μαρίτα Ουλσφογκ από την Επιτροπή Απασχόλησης ε, αναλαμβάνει την Προεδρία. Order, order. I'll give the floor to Ulrike. Ησυχία παρακαλώ. Ulrike Terebesius από την ECR. Έχετε το λόγο. Κυρία Κατάινεν, με όσο μας είπατε γραπτός, θα ασχοληθείτε ιδιαίτερα με τη μείωση της ανεργίας εντός της Ευρωζώνης ε, ενισχύοντας την κινητικότητα των εργαζομένων. Εγώ θα ήθελα να γνωρίσω από εσάς τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετανάστευση των εκπαιδευμένων νέων από την Νότια και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Δεν βλέπετε έναν κίνδυνο της λεγόμενης διαρροής εγκεφάλων που θα μειώσει την ανταγωνιστικότητα αυτών των χωρών. Και τι θα κάνουν οι χώρες που είναι ε, στόχος αυτής της κινητικότητας. Τι θα γίνει με διαφορετικό επίπεδο ε, και προδιαγραφές εκπαίδευσης ε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να έχουμε περαιτέρω εναρμόνιση και τελικά να πέσουν ξανά οι προδιαγραφές όπως έγινε με την Μπολόνια και θα ήθελα να σας πω ε, υπάρχει κάποια σκέψη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μαθαίνουν να καταργήσετε το επιτυχημένο σύστημα μαθητείας που έχουμε στη Γερμανία. Thank you. Σας ευχαριστώ. Κυρία Τρεμπέσιος, ξέρω πως κάποιοι, ή μάλλον έχω κάποιους φίλους, ιδιαίτερα στην Νότια Ευρώπη, που χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τη χώρα τους διότι δεν είχαν δουλειά. Κατά αυτή την έννοια, η ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων είναι λυπηρή γιατί αναγκάζονται να φύγουν από τη χώρα τους ε, επειδή δεν έχουν δουλειά. Ευτυχώς υπάρχει δυνατότητα να βρουν δουλειά αλλού στις, ε, στην Ευρώπη. Αλλά καταλαβαίνω αυτό που λέτε ότι η διαρροή εγκεφάλων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και να φεύγουν όλοι από τη χώρα. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να μπορέσουμε να εργαστούμε σε διάφορα επίπεδα για να αντιμετωπίσουμε την ανεργία των νέων. Η εγγύηση για τους νέους είναι ένα από τα μέσα. Και μπορούμε σταδιακά να επιταχύνουμε εδώ στο ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή τη διαδικασία, αλλά πρέπει να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε παρόμοια μέσα και σε διεθνές επίπεδο. Εμείς με την δικιά μου κυβέρνηση το φτιάξαμε αυτό το μέσο γιατί και μπορείτε να φανταστείτε ότι είμαι πολύ περήφανος γιατί ε, τώρα έχει αυτό αντιγραφεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, και να χαιρετήσω με την ευκαιρία και τους συναδέλφους που το προετοίμασαν ε, να αναφέρω δε και τη δυνατότητα να εναρμονιστούν τις να αναρμονιστεί η ποιότητα της εκπαίδευσης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια προϋπόθεση για το ότι ε, ε, τα διπλώματα και τα πτυχία σε μια χώρα να μπορούν να είναι αποδεκτά σε όλες. Ε, και είναι ένας, μια βασική προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει και η Μάριαν Χάρκιν από την Άλντε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, Υποψήφιοι Επίτροπε, καλώς ορίσατε. Χτες ε, η Είδαμε ότι στην έρευνα που ανακοινώθηκε ότι το εισόδημα που μπορεί κάθε νοικοκυριό να δαπανίσει ε, μειώνεται. Έχουμε δεν πέσει κάτω από το 4% για το 2015 και 2016 όσον αφορά την ανάπτυξη αυτού του εισοδήματος. Ε, εσείς μιλήσατε για τη ζήτηση, αλλά η ζήτηση χωλαίνει το δούνο του στην παγκόσμια εικόνα, οικονομική εικόνα δίνει, ε, λέει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση της ζήτησης όσο είναι μεγάλη η ανεργία. Γιατί και θα πει ότι τα κίνητρα θα δοθούν μόνο από την δανεισμό και όχι από την αύξηση των φόρων. Εσείς τώρα μιλήσατε για επενδύσεις χωρίς να δημιουργηθούν νέα χρέη. Πώς μπορούμε να μείνουμε ε, με αυτές τις δημόσιες επενδύσεις χωρίς να δημιουργηθεί νέο χρέος και έπειτα μιλήσατε για επενδύσεις και ανάπτυξη, αλλά είναι σαν το αυγό και την κότα. Ποιος ήταν πρώτος από τα δύο. Ευχαριστώ κυρία Χάρκιν. Είπατε ότι είναι σαν το αυγό του Κολόμβου, ναι. Καταρχήν πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει σταθερότητα και άρα χρειαζόμαστε επενδύσεις. Και εγώ πιστεύω ότι από αυτό θα, προέλθουν, προέλθει και η ε, ανάπτυξη. Τώρα, τα δημόσια χρήματα τα αρχικά δημόσια χρήματα ε, για επενδύσεις μπορούν να προέρθουν από πολλές και διάφορες πηγές. Καταρχήν, οι χώρες οι οποίες έχουν αυτή τη στιγμή πλεόνασμα θα μπορούσαν να επενδύσουν για το μέλλον και κάνοντας αυτό θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν και την οικονομία της Ένωσης. Θα πρέπει να υπάρξει συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση. Έχουμε κάποια πείρα από κάτι τέτοιο για να εξασφαλίσουμε ότι οι δημόσιες επενδύσεις δεν θα σημάνουν συγκέντρωση ελλείμματος και χρέους, γιατί ένα διαρκώς αυξανόμενο χρέος θα θέσει σε κίνδυνο την ανάκαμψη. Δεν θέλουμε να, πάρουμε, να αναλάβουμε άλλον κίνδυνο να δυναμητήσουμε την ανάκαμψη λόγω ψηλότερου δημόσιου χρέους. Όπως είπε και η Κρυσταλίνα την περασμένη εβδομάδα εδώ, αν δεν χρησιμοποιήσουμε πολλαπλασιαστές, αν δεν χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, δεν θα πετύχουμε πολλά καλύτερα. Και εδώ χρειαζόμαστε τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να είμαστε επίσης πολύ σταθεροί προς τα κρατη μέλη. γιατί χρειαζόμαστε και τη δική της ε, των κρατών μελών. Μαζί με το, την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να πείσουμε τα κράτη ότι χρειαζόμαστε ε, ε, τη χρήματα του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού και έπειτα αυξανόμενη ε, δυνατότητα δανεισμού της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή του EIF και των άλλων ε, τραπεζών. Ευχαριστώ πολύ. Oh, Όχι στην κυρία Χαρκίν, ο Μιγγέλ Βιέγκας από την ΚΟΕ. Ναι, κύριε, κύριε Κατάινεν, Πολύ με συγκίνησε ε, η εισήγησή σας. Εμείς στην Πορτογαλία είχαμε μια παρόμοια περίπτωση με τον Ντουράο Μπαρόζο, ο οποίος ε, διέφυγε για την Κομισιόν και άφησε σύξυλη την Πορτογαλία. Ε, γι' αυτό και καταλαβαίνω απόλυτα την παρέμβασή σας. Και θα ήθελα γι' αυτό Ωστόσο, να σας επιστήσω την προσοχή στη, στα όσα περάσαμε, στην εμπειρία μας. Τα, οι χώρες με τις περισσότερες ε, δημόσιες δαπάνες είναι αυτές που καλύτερα ε, αντιστάθηκαν στην κρίση και που ταυτόχρονα ε, δείχνουν καλύτερο δίκτυο κατανομής του πλούτου και, και του πλουτισμού. Η Φιλανδία, όπως ο ίδιος γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι από τις χώρες όπου υπάρχει πλούτος ε, και αντιστέκεται στην κρίση. Ενώ διαφορετικά στις υπόλοιπες χώρες υπάρχει μια πολιτική συγκέντρωση του πλούτου. Αν δεν μπορέσουμε να αντιστρέψουμε την πολιτική αυτή και να προωθήσουμε μια άλλη πολιτική που θα αξιοποιεί τους μισθούς, δηλαδή αντί να περιορίζονται οι φόροι στις επιχειρήσεις όπως έκανε η Φιλανδία, να, να, αφήσουμε, να αφήσουν τις συναλλαγές στο χρηματιστήριο. Κύριε Βιέγα, σας ευχαριστώ πολύ. Η ερώτησή σας αφορούσε το κατά πόσο θα πρέπει να έχουμε πιο σταθερή πιο σταθερά ε, εισοδήματα και μήπως θα έπρεπε να αυξάνουμε τους μισθού αντί να περιορίζουμε τους φόρους ε, των επιχειρήσεων. Ναι, όντως, εγώ ήμουν πρωθυπουργό σε μια πολύ ευημερή κοινωνία του κόσμου και η εικόνα που έχω για τον κόσμο από εκεί προέρχεται. Η ισότητα στη δικιά μας κοινωνία είναι βασική αξία. Επίσης δεν υπάρχει ούτε ένα κόμμα στη χώρα μου το οποίο να προτείνει την μείωση της βασικής, ε, του βασικού κράτους προνοίας. Σύμφωνα με τη δική μου εμπειρία, και δεν σημαίνει ότι όλοι συμμερίζονται αυτήν, ο ισχυρότερος εταίρος για μια καθολική κοινωνία πρόνοιας είναι η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, γιατί σε μια χώρα 500 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου ο δημόσιος τομέας παίζει πάνω από το 50% του ρόλου για το σύνολο της οικονομίας, η χώρα δεν θα μπορούσε να αντέξει ε, να έχει ένα από τα καλύτερα συστήματα ε, παιδείας ε, και, κοινωνικό, και κοινωνικής πρόνοιας, εάν δεν ήταν και από τις πιο ευημερούσες στον κόσμο. Χρειάζονται χρήματα δηλαδή και ελπίζω πως το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και η κοινωνική οικονομία της αγοράς θα βασίζεται σε, σε θέσεις υψηλής ποιότητας, σε ανώτατα εκπαίδευση, στην έρευνα και την, την ανάπτυξη ε, και σε ευέλικτη, ανοιχτή εσωτερική αγορά που δίνει την ευκαιρία στις παραδοσιακές βιομηχανίες αλλά και στις νέες startups. Η Τζιν Λάμπερτ των Πρασίνων. Σας ευχαριστώ. Με χαρά άκουσα στην ε, εισήγησή σας μια αναφορά στο κλίμα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί πιστεύουμε ότι το χαρτοφυλάκιό σας έχει εδώ ένα μέγα κενό και δεν αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι το κλίμα, η οικονομική και η κοινωνική κρίση δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν χωριστά. Η στρατηγική 2020 αναγνωρίζει ότι χρειάζεται αλλαγή στην πορεία και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση αλλά και για επενδυτικέ συμβάσει. Ποιε δράσει θα χρησιμοποιήσετε για να προωθήσετε αυτή την πράσινη μετάβαση ε, εντό τη Κομισιόν του Συμβουλίου και με του κοινωνικού εταίρου ώστε να δούμε κάποια πρόοδο και όχι απλά λόγια, ωραία λόγια. Ευχαριστώ. Υπάρχουν πολλά ε, που πρέπει να γίνουν και ο καθένας έχει τις δικές του μανίες. Μία από τις δικές μου είναι οι ανανεώσιμες και ανακυκλώσιμες πηγές ενέργειας από το τομείς εκτός του τομέα των τροφίμων. Εδώ πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο. Πρέπει να πω ότι δεν είμαι πολύ αισιόδοξο όταν βλέπω τις προτάσεις για πράσινη φορολογία που έχει υποβάλει η Κομισιόν για τα κράτη-μέλη δεν είναι και τόσο πρόθυμα να χρησιμοποιήσουν τα πιο καλά και τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για να προωθηθούν οι ανανεώσιμες ενέργειες και να δοθούν κίνητρα στις καλύτερες και πιο καθαρές τεχνολογίες, αλλά ε, θα, θα ε, συνεργαστώ με τον ε, με τους επιτρόπους που ασχολούνται με αυτού του τομεί, γιατί εγώ δημιούργησα νομοθεσία ε, για την ενέργεια ε, και λειτουργήσε από την πρώτη μέρα η μείωση των εκπομπών ε, ήταν πραγματικότητα. Επίσης το ίδιο είδος φορολογίες κάναμε και για τα αυτοκίνητα. Και αυτό είναι βέβαια ένα από τα θέματα και φυσικά το, η μεταρρύθμιση του συστήματος ανταλλαγής εκπομπών θα είναι πολύ σημαντική. Και αυτό είναι στην ατζέντα της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Πάτρικο Φλίν από την ομάδα FDD. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κατάινεν, ε, ο υποψήφιος επίτροπος Χιλ ε, δεν ήταν πρόθυμος να πει ότι θα προστατεύσει τα θεμητά συμφέροντα του City του Λονδίνου. Εσείς που είστε κατά κάποιο τρόπο το αφεντικό το αναγνωρίζετε ότι υπάρχει πλεονέκτημα σε ολόκληρη την Ένωση να έχουμε το, το πρώτο οικονομικό κέντρο του κόσμου εντός των συνόρων μας ή θα θέλατε ένα διαφορετικό Ευρωπαϊκό Σύνολο Οικονομικών Κέντρων με τη Φραγκφούρτη, για παράδειγμα, που ενθαρρύνεται να αναπτυχθεί για να περιορίσει την κυριαρχία του Λονδίνου. Σας ευχαριστώ. Για μένα, το πιο σημαντικό είναι ότι θα μπορούσαμε να διαφοροποιήσουμε ε, την αγορά κεφαλαίων μας, ώστε τα χρήματα να πηγαίνουν εκεί που χρειάζονται. Για μένα δεν είναι γεωγραφικό το ζήτημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είναι, μάλλον είμαι ευχαριστημένο αν αναπτύσσετε το Λονδίνο, αν αναπτύσσετε τη Φραγκφούρτη, αν αναπτύσσετε το Παρίσι ως οικονομικά κέντρα. Αλλά αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο είναι καλύτερη ένωση ε, αγορών, πράγμα το οποίο σημαίνει διάφορα πράγματα. Καταρχήν, να είναι πιο ελεύθερη η ροή κεφαλαίων από χώρα σε χώρα. Σημαίνει δημιουργία καλύτερων μέσων χρηματοδότησης, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η πρώτη ενέργεια που θα χρειαστεί να γίνει αν ε, μπορέσει να ξεκινήσει γρήγορα η Κομισιόν και αν επιβεβαιωθούμε εγώ και ο κύριος Χίλ είναι να αναπτύξουμε στάνταρ για ασφαλή τιτλοποίηση ή αποτιτλοποίηση για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το είδος το όχημα για να μπορέσουμε να έχουμε χρηματοδότηση μέσω αυτού. Έπειτα, για συνοριακές πληροφορίες πίστοσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και πάλι θέλουμε εδώ να τις βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες και τέλος να διευκολύνουμε την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς. για τις ιδιωτικές ε, επενδύσεις. Όπως σας είπα, πρόκειται για συγκεκριμένες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις μας να έχουν τη χρηματοδότηση και να έτσι με τη σειρά τους να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Ευχαριστώ. Ο Νίκολας Μπέιτς από τους μη εγγεγραμμένους. Έχετε το λόγο. Κύριε Επίτροπε, η λειτουργία και οι πολιτικοί προσανατολισμοί τη σήμερα δείχνουν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση τυφλώνεται από έναν ε, ε, φανατισμό του φιλελευθερισμού. Πριν από λίγα χρόνια με τη συνθήκη του Άμστερνταμ τροποποιήθηκε το άρθρο 42 της, της συνθήκης της Ρώμης που εννοούσε μια ελεύθερη ε, ανταλλαγή ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Πρέπει να επανέλθουμε εδώ για να ε, δώσουμε και πάλι νόημα στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Όμως στις απαντήσεις σας βλέπω τις ίδια, τα ίδια προβλήματα να εξακολουθούν να υπάρχουν. Θα δοθεί ε, προτεραιότητα στον εξυγχρονισμό της νομοθεσίας για την προστασία της απασχόλησης. Δηλαδή, στην ουσία δεν σημαίνει αυτό ακόμα πιο επισφαλή θέση των εργαζόμενων στην Ήπειρό μας. Αφού ούτω ή άλλω ευθυγραμμιζόμαστε με τη ΣΥΠΑ, γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε τα, μέσα, τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη αποδειχτεί λειτουργικά στη ΣΥΠΑ, γιατί να μην κάνουμε ένα ε, ε, άκτα όπως αυτό που έφτιαξε ο πρόεδρος Ρούσβελτ. Να αλλάξουμε δηλαδή όπλο, να προστατεύσουμε και εμείς τις επιχειρήσεις μας και τις θέσεις απασχόλησης που απειλούνται από την διεθνή ανταγωνισμό. Κύριε Κατάινεν. Ευχαριστώ. Συμφωνώ μαζί σας ως προς το ότι δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε ε, τους Κινέζους. Υπάρχουν και πολλές άλλες χώρες Υπάρχουν και άλλες χώρες στις οποίες δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε ως προς το επίπεδο του, των μισθών γιατί έχουν πολύ χαμηλούς ε, ε, μισθούς. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο βασίζεται σε άλλες αξίες και προοπτικές. Μιλάμε για ίσες ευκαιρίες για όλους και εργατικό δυναμικό με υψηλές δεξιότητες, γιατί χρειαζόμαστε προστιθέμενη αξία εκπαίδευση, έρευνα και εδώ χρειαζόμαστε προστιθέμενη αξία. Η Ευρώπη έχει πολλές χώρες που έχουν υψηλό επίπεδο ικανοτήτων, όπου δεν μπορούμε να έχουμε μία μαζική ε, παραγωγή και δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε το χαμηλότερο επίπεδο, με το χαμηλότερο επίπεδο μισθοδοσίας. Αυτό που έχει σημασία είναι οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς και αυτό αφορά και το εργατικό δυναμικό που πρέπει να βρίσκεται σε σωστά επίπεδα. Νομίζω ότι θα χάναμε πολύ περισσότερα εάν δεν είχαμε μια καλή συμφωνία με τις ΗΠΑ για το εμπόριο. Και από την άλλη πλευρά θα μπορούσαμε να κερδίσουμε ε, θέσεις εργασίας ε, με υψηλές δεξιότητες και προσόντα εάν ε, επιτύχουμε μια πολύ καλή εμπορική συμφωνία με τις Ιπα. Ο κύριος Κάσα από το ΕΛΚ. Από το παρελθόν μέχρι τώρα έπρεπε να προωθήσουμε μια πολιτική λιτότητας για να αντιμετωπίσουμε την κρίση στην Ευρώπη. Σήμερα λέμε ότι χρειαζόμαστε μια νέα πολιτική ως προς τις επενδύσεις, μια νέα επενδυτική πολιτική και ελπίζω να υπάρξει συμφωνία από όλες τις πολιτικές ε, ομάδες ως προς αυτό. Ακούσαμε για το επενδυτικό πακέτο των 300 δις. Εάν ε, γίνει αποδεκτό θα πρέπει να μας ορίσει η Κομισιόν τις προτεραιότητες και πώς θα πρέπει να δαπανηθούν αυτά τα χρήματα. Θα ήθελα να μου πείτε ποιες, ε, πώς ορίζονται αυτές οι προτεραιότητες και πώς μπορούμε να, χρησιμοποιήσουμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας που τόσο πολύ χρειαζόμαστε απάντηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κάσα. Οι προτεραιότητες λοιπόν. Θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και στη ζήτηση και στην προσφορά. Γιατί χρειαζόμαστε και τα δύο σκέλη για να επενδύσει ο ιδιωτικός τομέας. Επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους δημόσιους πόρους κατά τον πιο αποδοτικό τρόπο και είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε ε, νέο δημόσιο χρήμα και πόρους για να ανταποκριθούμε. Έτσι θα ξεκινήσουμε την πορεία μας. Θα χρησιμοποιήσουμε τον κοινοτικό προϋπολογισμό πιο αποτελεσματικά. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δημόσια, ε, δημοσιονομικά μέσα καλύτερα και θα ζητήσουμε από τις χώρες να επενδύσουν ε, στο μέλλον, ιδιαίτερα ως προς την έρευνα και την ανάπτυξη, αλλά και τις υποδομές. Θα ήθελα όμως να τονίσω ορισμένες προτερότητες από πλευράς ε, προσφοράς. Θα πρέπει να εφαρμοστεί σωστά το, ε, η οδηγία, η σχετική οδηγία και αν δείτε αυτό το γράφημα σε σχέση με την ανάπτυξη και την έρευνα θα δείτε ότι στην ψηφική αγορά ε, μιλάμε για 240 εκατομμύρια. 60 δις TTIP, ε, ε, ολοκλήρωση εσωτερικής αγοράς 60 δις. Πρόκειται για ένα χάρτη ευκαιριών. Σημαίνει ότι η Επιτροπή χρειάζεται πιο συντονισμένη δράση έτσι ώστε να νομοθετήσει και χρειάζεται τη δική σας υποστήριξη. Υπάρχουν ευκαιρίες. Δεν είμαι καθόλου απεσιόδοξος. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συλλέξουμε τις καλές μας ιδέες και να επικεντρωθούμε σε αυτά που μας ενώνουν. Ούτε Ούλμαν από τους ε, σοσιαλιστές και δημοκράτες. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, το πραγματικό έλλειμμα επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 200 δισεκατομμύρια το έτος και μετά το είπε και ο κύριος Γιουνκέρ, το είπατε και εσείς σας υποσχόμαστε ένα πρόγραμμα επενδύσεων 300 δισεκατομμυρίων για τα επόμενα χρόνια. Διαπιστώνω πως υπάρχουν δύο ομάδες ανθρώπων ε, ως προς την αντίδραση. Οι άλλοι λένε, οι μεν λένε πως ε, όχι δεν γίνεται και τα λέτε ψέματα αυτά μόνο και μόνο για να σας εγκρίνουμε και στην πραγματικότητα θα είναι κάτι σαν το σύμφωνο ανάπτυξη του κύριου Μπαρόζο. Άλλοι λένε πριν μάθουν καν ακριβώ τι είναι, πως είμαστε εναντίον. Εγώ σας κάνω μία πρόταση. Ελάτε πριν το τέλο του έτους στο Κοινοβούλιο, στις Επιτροπές, παρουσιάστε το πακέτο και ζητήστε να ψηφίσει το Κοινοβούλιο για αυτό το πακέτο είστε διατεθειμένος για κάτι τέτοιο ή για όχι. Αναφερθήκατε πολλές φορές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ζητήσατε τη βοήθειά μας, θέλετε ε, να υπάρξει μια τέτοια σοφορία ή όχι. Για μένα είναι σημαντικό αυτό το ερώτημα για την αξιολόγηση της Κομισιόν. Thank you. Mr. Σας ευχαριστώ κύριε Μπούλμαν. Το... Η ερώτησή σας ε, βεβαίως ήταν ότι ασχολούμαι με αυτό το θέμα μόνο και μόνο γιατί θέλω να γίνω επιτροπός. Όχι, είμαι πολλά χρόνια ε, πολιτικός και είμαι πολιτικός γιατί θέλω να αλλάξω τον κόσμο. Προσπαθώ να φτιάξω μια καλύτερη Ευρώπη από διάφορες θέσεις και ακόμα και τώρα παρετήθηκα από Πρωθυπουργός για να γίνω Επίτροπος για να δημιουργήσω μια καλύτερη Ευρώπη. Αυτή είναι η πρόθεσή μου και ευχαρίστω εάν το δεχτεί το Κοινοβούλιο θα ήθελα να συνεργαστώ για τα θέματα των επενδύσεων της ανταγωνιστικότητας και των θέσεων εργασίας. Αν μου επιτρέπετε τώρα να αναφερθώ στο εξή εγώ θα προσπαθήσω βεβαίως να οργανωθούμε καλύτερα αν για να μπορέσω να απευθυνθώ στο κοινοβούλιο ακριβώς για να δούμε Ποιε θεωρείτε εσείς ότι είναι οι αποτελεσματικότερε επενδύσεις. Βεβαίως δεν υπάρχει ακόμα η νέα επιτροπή, αλλά ανάλογα με τις αποφάσεις σα θα ήθελα και εγώ πράγματι να οργανώσουμε ε, τέτοιες ημερίδες έτσι ώστε διάφοροι επίτροποι και εγώ να έρθουμε να συναντήσουμε τους ε, βουλευτές και να ακούσουμε τι απόψει σα. γιατί αναφέρεται πράγματι και τις διαφορετικές ε, γεωγραφικές στοιχείες. Έχω ακόμα 10 δευτερόλεπτα. Θέλω μία απάντηση για την ψηφοφορία. Όταν μιλάμε για λεφτά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέλω να μου απαντήσετε σας παρακαλώ κύριε υποψήφιο επιτροπέ. Εάν κατάλαβα καλά, και δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβα καλά. Ε, θα συνεργαστώ με την Κρυσταλίνα Γεωργίευα για να χρησιμοποιήσουμε τον κοινό μας προϋπολογισμό πιο αποτελεσματικά ακριβώς για να ε, έχουμε μια μόχλευση για επενδύσεις. Ταυτόχρονα, όταν μιλάμε για νέα ορμή και νέα κονδύλια, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά τα χρήματα των φορολογουμένων για να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας. Ευχαριστώ. Hans Olaf Henkel από το ECR έχετε τον λόγο. Κύριε Κατάινεν, στο χαρτοφυλακείο σας υπάρχει η λέξη ανταγωνιστικότητα. Πριν από πολλά χρόνια υπήρχε ένας επίτροπος, ο Λέων Μπρίταν, που πάντα ε, ρωτούσε το εξή θα γίνει ανταγωνιστική η Ευρώπη και απαντούσε με τον ανταγωνισμό. Η Κομισιόν όμως ε, ζητάει ακριβώς το αντίθετο και είναι υπέρ της εναρμόνισης. Ο Επίτροπος Άντορ ζητάει ένα κοινό σύστημα ανεργίας, ε, επιδόματος ανεργίας. Αντί για φορολογικό ανταγωνισμό η Κομισιόν τώρα θέλει φορολογική εναρμόνιση. Ο πρόεδρος Γιούνκερ θέλει ευρωομόλογα και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση δεν είναι παρά κοινωνικοποίηση των εθνικών τραπεζικών ρίσκων. Μπορεί έτσι να σταθεροποιηθεί προσωρινά το ευρώ, αλλά εγώ θα σας ρωτήσω κάτι το απλό. Τι θεωρείτε ότι κάνει αυτή η εναρμόνιση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο. Κύριε Χένκελ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ερώτημά σας αφορούσε την εναρμόνιση και το εάν βοηθάει ή όχι ή εάν δημιουργεί κάποιες ε, τεχνητές δομές που δεν βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα. Η εναρμόνιση για εμένα σημαίνει πως ε, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες και οι ίδιες συνθήκες για όλους. Οπότε θα πρέπει να έχουμε ίσους όρους ανταγωνισμού. Ταυτόχρονα, εναρμόνιση δεν σημαίνει πως ε, ταιριάζουν τα ίδια σε όλους. Και βεβαίως ε, πρέπει να διαλέξουμε πάρα πολύ προσεκτικά τους τομείς στους οποίους χρειαζόμαστε εναρμόνιση και ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους δεν χρειαζόμαστε περαιτέρω εναρμόνιση. Αυτό είναι ένα ερώτημα επικουρικότητας. Οπότε εγώ θεωρώ πως υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα στα οποία χρειαζόμαστε πιο εναρμονισμένη πολιτική. Παραδείγματο χάρη η ενιαία αγορά. Η Ενιαία αγορά ενέργειας παραδείγματο χάρη. Ή η αυστηρή εφαρμογή της οδηγίας ε, υπηρεσιών. Αυτά είναι τα μέτρα στα οποία χρειαζόμαστε περισσότερη εναρμόνιση. Ταυτόχρονα υπάρχουν πολλά θέματα στα οποία είναι καλύτερο το τοπικό ή το εθνικό επίπεδο, γιατί είναι πιο αποτελεσματικό και δεν θα έχει, νομίζω, επιβλαβείς επιπτώσεις. Σας ευχαριστώ. Ντομινίκ Ρικέ από την ομάδα Άλντε έχετε το λόγο. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, χρειαζόμαστε χρηματοδότηση και μιλάμε για ένα ε, δις. Ε, υπάρχουν ε, πολλά ελλείμματα και στα διαρθρωτικά ταμεία. Ο μηχανισμός Connecting Europe έχει μόνο 33 δις και δυστυχώς τα ιδιωτικά κεφάλαια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις υποδομές. Όλοι αναρωτιόμαστε πού θα βρεθούν τα 300 δις που αναζητά ο πρόεδρος Γιούνκερ. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω τα εξής. Θα είσαστε ε, υπέρ ε, αμοιβαίων κεφαλαίων που θα πρέπει να βασίζονται στα στοιχεία, στα στοιχεία ενεργητικού που διαθέτουμε και επίσης θα χρησιμοποιήσετε ρυθμιστικά μέσα για τα ιδιωτικά κεφάλαια τα οποία να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν σε δημόσια επενδυτικά έργα. απάντηση. Κύριε Ρικέ, σας ευχαριστώ. Το ερώτημά σας αφορά την χρηματοδότηση των μεγάλων προγραμμάτων υποδομών. Και μας ενδιαφέρει να ξέρουμε από πού θα προέλθουν αυτά τα χρήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα είναι ένα από τα δύσκολα θέματα του μελλοντικού μου χαρτοφυλακίου. Πρόκειται για ένα τομέα που με απασχολεί ιδιαίτερα, δηλαδή οι μεταφορές. Θα πρέπει να βρούμε τρόπο για νέα καινοτόμα προγράμματα και ευκαιρίες. Πιστεύω ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα πρέπει να προσελκύσουν ε, ιδιωτικό χρήμα. Ε, τα 300 δις δεν είναι μόνο ε, ρευστό. Θα χρησιμοποιηθούν και άλλα ρυθμιστικά μέσα έτσι ώστε να φτάσουμε στα 300 δις το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη τώρα. Ε, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ομολογίες έργου πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Είχαμε ορισμένες καλές εμπειρίες από ομολογίες έργου, ακόμα και σε πιλωτικά προγράμματα. Νομίζω όμως ότι θα διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο, ιδιαίτερα σε έργα ε, υποδομών. Η Φερεγγιότητα 2 και η κεφαλιακή αγορά θα μας βοηθήσουν καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Και αυτό θα μας απασχολήσει με τον ε, Τζόναθαν Χιλ. Λίν Μπόλεν από την Γκουέ. Ευχαριστώ. Η ανεργία στην Ιρλανδία παραμένει μεγάλο πρόβλημα και 250.000 έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Τώρα ο δείκτης ανεργίας ανέρχεται σε 23%. Τα τελευταία χρόνια έχει ε, μειωθεί η δημόσια, οι δημόσιες, έχουν μειωθεί οι δημόσιες επενδύσεις και νομίζω ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε της, ε, την οθρή πολιτική του, της ΕΚΤ που οδήγησε σε αυτή την κρίση και στο ανακοινωθέν τύπου του Συμβουλίου Υπουργών στο 2012, 12, με συγχωρείτε, όρισε ότι το σχέδιο διάσωσης θα πρέπει να οδηγήσει σε επανακεφαλαιοποίηση. Άρα η ερώτησή μου είναι αναθεωρήσατε τη θέση σας και εάν όχι μπορείτε να μας πείτε πώς μπορεί να επενδύσει δημόσια ε, η Ιρλανδία για θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα για τους νέους τη στιγμή που η Ιρλανδία καλείται να διασώσει το ευρώ. Ευχαριστώ κυρία Μπόρεν. Η ερώτησή σας σχετίζεται με το πώς μπορεί κανείς να επενδύσει σε θέσεις εργασίας και απασχόληση, γιατί η Ιρλανδία ε, λαμβάνει μέτρα, ε, ρυθμιστικά μέτρα και οι Ιρλανδοί βρίσκονται σε πολύ δυσχερή θέση. Κατανοώ την θέση των Ιρλανδών πολιτών και θα πρέπει να πω ότι οι Ιρλανδοί είναι ε, ιδιαίτερα θαραλέοι και αναλαμβάνουν την ευθύνη των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα. Η Ιρλανδία είναι μία από τις χώρες Ε, όπου πιστεύω ότι θα ε, υπάρξουν πολλές ιδιωτικές επενδύσεις, διότι η Ιρλανδία αντιμετωπίζει τις δικές υποθέσεις μόνη της, παρόλο που είναι δύσκολο. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε κοινά ευρωπαϊκά ε, μέτρα. Θα πρέπει πρέπει τα διαρθρωτικά ταμεία να χρησιμοποιούνται καλύτερα, να βρεθούν νέα ε, χρηματοοικονομικά μέσα για την χρηματοδότηση των έργων υποδομών και να δώσουμε βάρος στην έρευνα και την ανάπτυξη. Όλα τα κράτη βρίσκονται σε παρόμοια θέση. Ακόμα και οι πιο στεναρές χώρες δεν ξέρουν αν θα βρίσκονται στην ίδια θέση μετά από 10 χρόνια, γιατί θα πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις παντού για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Έρνεστ Ούρτασον από τους ε, Πράσινους υπέρμαχος της λιτότητας που απέτυχε. Πριν γίνεται επίτροπος, το 2010 είχατε ταχθεί ε, κατά των ευρωομολόγων και τον Ιούλιο μιλήσατε υπέρ της ε, Τρόικας λέγοντας ότι είναι υπέρμαχος των χωρών πιστωτών. Νομίζω ότι κύριε Κατάινεν ε, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι με τις επενδύσεις δεν έχει γίνει τίποτα. Πείτε μας κάτι για το δημόσιο χρήμα που ε, εντάσσεται στα πολυετή μας προγράμματα. Πείτε μας πώς θα οριστεί το επενδυτικό πρόγραμμα της Επιτροπής. Πείτε μας κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο, γιατί μέχρι τώρα δεν το κάνατε. Πώς Εσείς είπατε ότι τάχθηκα κατά του πακέτου της Ελλάδας και της Πορτογαλίας. και από πού πρέπει να προέλθουν τα χρήματα για τις επενδύσεις. Εγώ ήμουνα υπέρ και των δύο πακέτων για την Ελλάδα. Ε, αντίθετα με μερικούς άλλους από τη χώρα μου και ως υπουργό Οικονομικών. Προσπάθησα να πείσω τους Φιλανδούς να δεχτούν το σχέδιο αρρωγής προς την Πορτογαλία και αυτό δεν ήταν καθόλου ε, δημοφιλές. Ως Πρωθυπουργό και υπουργό Οικονομικών κατέβαλα κάθε προσπάθεια για να συμμετάσχει η χώρα μου σε αυτά τα προγράμματα. Και για οικονομικούς λόγους, αλλά και λόγω αλληλεγγύης. Αλλά δεν ήταν καθόλου εύκολο οι Φιλανδοί που έχασαν τις εργασίες τους ε, εξαιτίας της κρίσης σε άλλα μέρη της Ευρώπης αναρωτήθηκαν γιατί να δανείσουμε χρήματα σε εκείνους που δημιούργησαν την ε, κρίση τη στιγμή που εμείς χάσαμε την εργασία μας. Αυτά έλεγαν πολλοί συμπολίτες μου. Ελπίζω να αρθούν αυτά τα χάσματα μεταξύ των λαών. Καταλαβαίνω ότι οι Έλληνες, οι Πορτογάλοι, οι Ιρλανδοί, οι Ισπανοί είναι πολύ απογοητευμένοι. Θα ήθελα να ε, φέρουμε τους ανθρώπους πιο κοντά. Αλλά νομίζω ότι ε, θα πρέπει τα χρήματα να προέλθουν από εκείνους που είναι πλεονασματικοί και να γίνει καλύτερη χρήση του κοινοτικού προϋπολογισμού. Χρειαζόμαστε και μια κοινή προσπάθεια από την Ευρώπη. Και τέλος θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να αποστείλουμε ένα ενθαρρυντικό μήνυμα προς τους πολίτες Ας μην αναμοχλεύουμε το παρελθόν και ας δούμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Thank you. Ε, ε, e Μάρκο Βάλε, από την Ευρώπη για τη Δημοκρατία και την Ελευθερία. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα σας. Μιλήσατε για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις μέσα στο πρόγραμμα των 300 εκατομμυρίων. Μιλήσατε για οικονομία αλλά για πολύ ευαίσθητα δημοσιονομικά μέσα. Αυτό πολύ μας ανησυχεί. Η οικονομία είναι 1-3, η πραγματική οικονομία 750 χιλιάδες ε, ε, εκατομμύρια. Εσείς θέλετε να κάνετε, ε, ε, να προστατεύσετε αυτή την μπάλα, αυτή τη σφαίρα. Έπειτα υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στην πραγματική οικονομία και την κοινωνία. Η οικονομία ήδη επηρεάζει πάρα πολύ υπερβολικά την πολιτική. Μα ζητάτε όμω θυσίε και μεταρρυθμίσει. Αυτό θα είναι το μπόνους για του ιδιώτε. ενώ σφίξιμο του ζωναριού και διαρθωτική φτώχεια θα σημάνει για του απλούς πολίτε τη Ευρώπη. Πρέπει ανοίξουμε πόρτες στους ιδιώτες επενδυτές μέσω από αυτά τα ε, μέσα. Μήπως πρέπει να ανοίξετε, να, δείτε ποια είναι η πραγματική οικονομία από αυτή την ε, εικονική ε, οικονομία. Ο κύριος Κατάινεν. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει όντω να δημιουργήσουμε τι προποθέσει για του μικρούς επενδυτέ, αυτού που έχουν ε, τα χρήματα για να αγοράσουν μετοχέ για ε, των εταιριών. Και πώς θα δημιουργήσουμε μια δίκαιη αγορά. Ε, μιλήσατε για τα πριμ των τραπεζικών Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπαρνιέ για τα όσα έχει κάνει σε αυτό το τομέα. Τώρα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη και η τραπεζική βιομηχανία ολόκληρη θα ακολουθήσει πραγματικά τους νέους κανόνες που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Και βέβαια η εφαρμογή της Τραπεζικής Ένωσης είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί είναι ο τρόπος για να αυξηθεί η σταθερότητα. Εξίσου θα πρέπει να προσέξουμε ε, την υψηλή ποιότητα τετλοποίηση, ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, να έχουν νέες ευκαιρίες για χρηματοδότηση. Υπάρχουν πολλά χρήματα στους ε, ιδιωτικά στην Ευρώπη, αλλά για κάποιους λόγους δεν πηγαίνουν εκεί που χρειάζονται περισσότερο. Για να μπορέσουμε λοιπόν να ενισχύσουμε την ευημερία και την ευμάρεια στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε κυρίω θέσει απασχόληση. Ο ιδιωτικό τομέα είναι αυτό που τι δημιουργεί και όχι οι κυβερνήσει ή τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία πολιτική που έχουμε και να δημιουργήσουμε καλύτερη ενιαία αγορά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για την παραδοσιακή βιομηχανία, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε και νέες θέσεις. From Γκροστέτ e από το Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Κατάινεν. Επανέρχομαι στη νέα στρατηγική για την ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αναμένεται για το 2015. Πώ μπορείτε να εγγυηθείτε ότι τα συγκεκριμένα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη στρατηγική δεν θα μείνουν νεκρό γράμμα θα μετα... και ότι θα μεταφραστούν σε πραγματικέ και συγκεκριμένε δράσει. Γιατί πέρα από τα μεγάλα σχέδια υπάρχει ένα μέγα δυναμικό ανάπτυξη το οποίο ε, δράζεται στην ε, εφαρμογή της ισχύουσα νομοθεσία. Πριν να υποβάλλετε νέες προτάσεις, σκοπεύετε να αξιολογήσετε τα αποτελέσματα και το δυναμικό της υπάρχουσας ε, νομοθεσίας, ε, μεταξύ άλλων στον τομέα της ενίας αγοράς. Και έπειτα για το μέγα αυτό πλάνο επενδύσεων 300 δις. Πολλά πρέπει ακόμα να γίνουν στον τομέα της ενέργειας και του ψηφιακού τομέα. Ποια μέτρα σκοπεύετε να λάβετε ώστε να εξασφαλίσετε τα κράτη-μέλη και οι τοπικές αρχές που σύγχανα. Ε, χρειάζονται τέτοια χρήματα θα είναι έτοιμες για να χρησιμοποιήσουν αυτό το, αυτό το νέο, τη νέα χρηματοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κοιτάξτε, ε, <laughs> πολύ περισσότερα από 300 δις χρειάζονται για αν θέλουμε να υπερασπιστούμε το κοινωνικό πρότυπο της Ευρώπης και να ενισχύσουμε την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Το μοντέλο μας θα πρέπει να βασίζεται σε βιώσιμες αξίες. Και εκεί ο ένας άξονας είναι οι θέσεις ψηλής ποιότητας. Αυτό λοιπόν θα το φροντίσουμε μαζί με τη Μαρία Τάισεν. Δεν μπορούμε να δεχτούμε το κοινωνικό ντάμπινγκ. Πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα και την ανάπτυξη. Πρέπει να κάνουμε μεταρρυθμίσεις σε εθνική σε εθνικέ ρυθμίσει για να υπάρξει ανάπτυξη και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα. Και σωστά είπατε ότι πρέπει να εφαρμόσουμε την ισχύουσα νομοθεσία και όσα μέσα έχουν ήδη ε, υιοθετηθεί. Η οδηγία για τις υπηρεσίες είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Αν λειτουργούσε και εφαρμοζόταν σωστά, θα είχαμε περισσότερες δουλειές στην Ευρώπη. Πιστεύω πως έχουμε φτάσει σε μια νέα φάση στην ευρωπαϊκή οικονομία. Και Όντως πρέπει να εστιάσουμε στις επενδύσεις για να δημιουργήσουμε κάτι νέο. Έχει επανέλθει η εμπιστοσύνη και έπειτα όμως θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, να χρησιμοποιήσουμε το χρήμα του ιδιωτικού τομέα, να δημιουργήσουμε καλύτερη νέα αγορά για να υπερασπιστούμε όλους τους τομείς, την ενέργεια, το ψηφιακό τομέα και να εφαρμόσουμε όλα τα άλλα μέτρα που έχουμε ήδη αποφασίσει. Και έπειτα οι πόροι του, δημόσιου τομέα θα πρέπει να, χρησιμοποιηθούν επίση πιο αποτελεσματικά. Η κυρία Μπερέση. Κύριε Κατάινεν, πιστεύω πως η Ευρώπη δεν θα είναι μια μεγάλη Γαλλία. Αλλά έχω την εντύπωση πως ε, πιστεύετε πως θα πρέπει να είναι μια μεγάλη Φιλανδία η Ευρώπη. Και επίσης ότι ξεχνάτε πως ακόμα και ο κύριος Βαρόζο είχε θεωρήσει που το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο ήταν ένα στοιχείο που ωφελούσε την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Όταν λοιπόν μας μιλάτε για την επιστροφή της εμπιστοσύνης, πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί τι πράγμα μου μιλάτε. 57% των Ευρωπαίων δεν συμμετείχαν στις τελευταίες ευρωεκλογές. Ίσως όμως εδώ να έχουμε ένα σημείο διαφωνίας. Εμένα αυτό δεν μου φαίνεται για επιστροφή της εμπιστοσύνης. Όταν ε, αναζητάτε το βασικά τα, τα, τα, βασικά στοιχεία για τα 300 δις που υποτίθεται είναι το βασικό εργαλείο για να ξανακερδίσετε την εμπιστοσύνη. Μα δεν μας πείτε τίποτα. Πώς θα κάνετε, πού θα τα βρείτε για να χρηματοδοτήσετε τις επενδύσεις ε, χωρίς να χρεωθείτε. Αν θέλετε ας πούμε να στηρίξετε το φόρο για τις συναλλαγματικές ε, τις, ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Υπάρχουν μέσα. Ίσως να βγάλετε ε, τις δαπάνες του Διευθυντικού Ταμείου και να αφαιρεθούν από το έλλειμμα. Είστε στο Ευρωκοινοβούλιο. Ποια είναι η δέσμευσή σας όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και ψήφο του Κοινοβουλίου για το σχέδιο αυτό επενδύσεων. Κύριε Κατάινεν, παρακαλώ. Euh, there were several Ευχαριστώ κυρία Μπερές. Ε, διάφορες πτυχές περιλάμβανε η ερώτησή σας που κάλυπταν τα συγκεκριμένα μέτρα ε, προγράμματα για το επενδυτικό πακέτο και κατά πόσο θα χρησιμοποιηθεί ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών ε, συναλλαγών και ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα. Όπως είπε ο πρόεδρος Γιούνκερ, θα πρέπει να, υπάρξει ένα συνολικό επενδυτικό πακέτο το οποίο θα εντοπιστεί εντός των πρώτων τριών μηνών της, ε, από τη σύσταση της Κομισιόν. Αυτό είναι η πολιτική κατευθυντήρια γραμμή που θα εφαρμόσουμε εάν ε, ε επιβεβαιωθώ στη θέση αυτή. Επίσης, έχουμε αρκετά καλά πει από πού θα προέρθουν τα δημόσια χρήματα για αυτό το πακέτο επενδύσεων. Μπορώ και να το επαναλάβω. Καλύτερη χρήση της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων μέσων ε, ευρωπαϊκών, ε, το καλύτερη χρήση των εθνικών επενδυτικών τραπεζών και καλύτερη χρήση του ευρωπαϊκού προπολογισμού ώστε να χρησιμοποιηθούν καλύτερα αυτοί οι πόροι που υπάρχουν αλλά και εθνικοί προπολογισμοί των κρατών που έχουν αυτή τη στιγμή πλεόνασμα. Έπειτα, συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όλες μας οι πολιτικές δεν θα αυξήσουν το έλλειμμα και το χρέος. Ελπίζω πως θα κατανοήσετε επίσης και δεν μπορώ να αποκαλύψω τα πάντα σε αυτή τη φάση, διότι ο πρόεδρος Γιούνκερ, όπως και εγώ, δεν έχουμε ακόμα μπορέσει να τα συζητήσουμε όλα σε όλες τις λεπτομέρειες με, όλους τους, με τους μελλοντικού μας συναδέλφους και επίσης ίσως κάποια μέτρα να χρειαστεί να συγκεντρώσουν ευρεία πολιτική συνένεση για να έχουν ευρύτερο αντίκτυπο, οπότε για να αποφύγουμε αρνητικές αντιδράσεις δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Παρακαλώ να τηρείτε πιο αυστηρά το χρόνο σας, διότι ε, είμαστε λίγο πίσω στο χρονοδιάγραμμα. Ο κύριος Κοτέρο από την CR. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, και καλωσορίσατε στην Επιτροπή μας, ε, κύριε Κατάινεν. Δύο ώρες ε, περίπου μιλάμε, αλλά ακόμα έχω την αίσθηση πως δεν έχω καταλάβει τι είναι το πρόγραμμα δράσης σας. Τι θα κάνετε στην ουσία, γιατί αν θέλετε να κερδίσετε την εμπιστοσύνη μας για τις ικανότητές σας, χρειαζόμαστε συγκεκριμένα παραδείγματα. Τι σκοπεύετε να κάνετε. Μας είπατε ότι... Ε, θα αναζητήσετε πιο καινοτόμε λύσει και ότι θα χρησιμοποιήσετε πιο αποτελεσματικά τα δημόσια χρήματα, καλύτερη χρήση των διορθωτικών ταμείων, είπατε, και τέτοια. Όμως συγκεκριμένα πώς θα χρησιμοποιήσετε καλύτερα τα δημόσια κονδύλια, πώς θα βρείτε πιο καινοτόμες λύσεις, ποιες είναι αυτές οι πιο καινοτόμες λύσεις. Δεν χρειάζεται να μακρηγορήσετε, αλλά να μας πείτε ξεκάθαρο κατάλογο δράσεων. Παρακαλώ, μη μας λέτε ποιες είναι οι καλές σας προθέσεις. Ξέρουμε ότι οι προθέσεις είναι καλές. τι θα κάνετε συγκεκριμένα. Κατάινεν, ευχαριστώ πάρα πολύ το ερώτημά σας. Τι είναι το τι θα κάνουμε συγκεκριμένα στο πακέτο των επενδύσεων. Πρώτα απ' όλα δεν είχα την ευκαιρία να έχω ανταλλαγή απόψεων ε, ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι σήμερα. Θα ήθελα να ακούσω τις δικές σας απόψεις για το ποια είναι τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία. Κατόπιν δεν είχα και την ευκαιρία να συνομιλήσω με τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και τους συναδέλφους επιτρόπους για το τι θα κάνουμε αν έχουμε τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Δεν είχα παραδείγματο χάρη ακόμα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τον Πιέρ πώς θα χρησιμοποιήσουμε το, ε, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή τη φορολογία για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Ελπίζω να αντιλαμβάνεστε πως δεν είναι τα πάντα έτοιμα γιατί ακόμα δεν έχει συσταθεί σε σώμα η Νέα Επιτροπή. Κάποια παραδείγματα όμω, η Κρυσταλίνα την προηγούμενη εβδομάδα είπε πώ θα ήθελε να διπλασιάσει το ποσό των επιχορηγήσεων από το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Έτσι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και εδώ πέρα συμφωνώ μαζί της. Επίσης, ε, για τα έργα, για τα ομόλογα έργου, πράγματα να τα χρησιμοποιήσουμε. Για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, θα έρθουμε σε συνεννόηση με τον πρόεδρο Χόιερ ακριβώς και για την ανεργία των νέων και για την εκπαίδευση που δεν υπάρχει ακόμα αρκετή εμπλοκή της τράπεζας. Επίσης θα συνεργαστώ στενό με τον πρώτο αντιπρόεδρο για να μειώσουμε την ανεργία και την ε, γραφειοκρατία και την υπερβολική ρύθμιση κτλ. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο κατάλογος, θα απαντήσω και στι επόμενε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ όλοι Ρεν από τους φιλελεύθερους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Υποψήφιο Επίτροπε, έχετε μια πάρα πολύ σημαντική, θα έχετε πάρα πολύ σημαντική δουλειά όσο Επίτροπος ο Αρμόδιος για την ανταγωνιστικότητα. Ε, η παραγωγή βιώσιμης ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Εξαρτώμεθα πάρα πολύ από τις, ε, τα ορυκτά καύσιμα και ε, ειδικά και από την Ρωσία. Το είπε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από λίγους μήνες όταν είπε πως θα πρέπει να βελτιωθεί η ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία και η δική μας η ε, ανθεκτικότητα απέναντι σε εξωτερικά σοκ. Ως Αντιπρόεδρος της Κομισιόν πώς θα διασφαλίσετε το ότι θα μειωθεί η εξάρτησή μας από εισαγόμενη ενέργεια ε, πώς θα στηρίξετε την ε, βιοενέργεια, πόσα από αυτά τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ θα αφιερώσετε για αυτό τον ε, σκοπό. Η βιώσιμη πράσινη οικονομία είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και από την πλευρά της περιφερειακής ανάπτυξης, ειδικά στην Ανατολική Φλανδία, την οποία γνωρίζουμε και οι δύο πάρα πολύ καλά. Σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση αυτή από τον προκατοχό μου, τον κύριο Ρέν. Το θέμα αυτό αφορά ακριβώς ε, την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη και το πώς θα έχουμε καθαρή πράσινη ενέργεια και ταυτόχρονα πώς θα αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Το πρώτο συγκεκριμένο εργαλείο είναι οι επενδύσεις στην ενέργεια, στις διασυνδέσεις, παραδείγματος χάρη στην Ιβυρική. Η Ισπανία και η Πορτογαλία πώς θα συνδεθούν με την ε, Γαλλία. Και η Φιλανδία επίσης ε, με τη διασύνδεση με τις βαλτικές χώρες και από εκεί με την υπόλοιπη Ευρώπη. Καμία περιοχή από τις δύο δεν πρέπει να παραμείνει ενεργητικά απομονωμένη. Και βεβαίως δεν πρέπει όσον αφορά τις εισαγωγές να είμαστε εξαρτημένοι από μία πηγή μόνο. Βεβαίως καμιά φορά ε, εξάγουμε και αέριο. Πρέπει λοιπόν να δούμε εδώ πέρα τι μπορεί να γίνει και με την έρευνα και την ανάπτυξη. Πιστεύω πάρα πολύ λοιπόν στις δυνατότητες που προσφέρει η ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας και οικονομίας. Μπορεί να βελτιωθεί και η κατάσταση της ανεργίας, να δημιουργήσουμε ανάπτυξη Υπάρχουν κάποια... κάποιες προστατευτικές ε, τάσεις ε, λοιπόν ε, που είναι κυρίως μη δασμολογικά εμπόδια όσον αφορά την εισαγωγή και εξαγωγή πράσινη ενέργεια. Σας ευχαριστώ. Είναι τώρα η σειρά μου να προεδρεύσω. Σας ευχαριστώ κυρία Όλυστοκ. Να σας πω από την αρχή πω έχουμε καθυστερήσει κατά δέκα λεπτά. Και λυπούμε βεβαίω γιατί έχουμε ακόμα 45 βουλευτές που πρέπει να θέσουν ερωτήσεις. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ευθυροί. Κυρία Παλώμα Λόπες. Κύριε Κατάινα, οι στόχοι ε, δημόσιας επένδυσης για την ε, Ευρωζώνη είναι χαμηλές και δεν μπορούμε να φέρουμε σε πέρας τις δημόσιες επενδύσεις, ενώ οι ιδιωτικές επενδύσεις δεν είναι επαρκείς. Η ΕΚΤ ασχολείται με τον έλεγχο των τιμών και όχι με την απασχόληση. Θα προωθήσετε τη βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση μπροστά ε, το, στο κοινωνικό dumping. Τι θα κάνετε για να εγγυηθείτε ότι, στο ότι οι επενδύσεις θα είναι πραγματικά παραγωγικές για όλα τα κράτη-μέλη. Θα καταπολεμηθεί η φορολογική απάτη ή θα συνεχίσετε με τις ε, τρέχουσες πολιτικές που δημιούργησαν μεγάλη ζημία. Ε, δεν θα πρέπει να διαβάζετε όμως και τόσο γρήγορα, διότι ίσως ανακύψουν προβλήματα όπως καταλαβαίνετε. Κύριε Υποψήφιο Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Παλώμα Λόπες για την ε, ερώτησή σας. Η πρώτη ερώτηση είναι κατά πόσο θα προωθήσω τα επενδυτικά πακέτα στο δημόσιο τομέα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η απάντησή μου είναι ε, θετική, είναι καταφατική. Το θεωρώ καθήκον μου και επίσης θα δημιουργήσω ευκαιρίες για να υπάρξουν και ιδιωτικές επενδύσεις. Υπάρχουν πολλά ε, θετικά στοιχεία στην Ευρώπη, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να προχωρήσει πάντα όπως θα θέλαμε. Ε, επίσης, πώς θα καταπολεμήσω το κοινωνικό ντάμπινγκ. Θα ήθελα να είμαι απόλυτα σαφής. Ε, η οικονομία της αγοράς και ε, όπως διαμορφώνεται ορίζει ότι δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνικό ντάμπινγκ, δεν έχει θέση στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι η οικονομία της αγοράς με βάση την ε, κοινωνική αυτή συνιστόσα είναι κάτι που μας βρίσκει ε, σύμφωνος. Ο πρόεδρος Γιούνκερ είπε ότι η οδηγία για τους αποσπασμένους θα πρέπει να εφαρμοστεί αυστηρά και θα συνεργαστώ με την Μαριάν ε, Τάισεν επί του θέματος με την ε, εφαρμογή της οδηγίας και εξετάζοντας την ίδια την οδηγία. Χρειαζόμαστε όμως ε, διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η κυρία ε, Μόνικα Βάνα από την Ρέτζη. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, μιλήσατε πάρα πολύ για τα οικονομικά μέσα, λιγότερο για τα ε, για τα διαρθρωτικά ταμεία. Αλλά βέβαια εξίσου σημαντική είναι και αυτή η πολιτική και η πολιτική περιφερειακή. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς ε, θα διατεθούν αυτά τα 300 δισεκατομμύρια. Ε, το ερώτημά μου λοιπόν είναι πώς ε, πόλεις και περιφέρειες έχουν ήδη προγραμματίσει ότι θα κάνουμε αυτά τα κονδύλια, π.χ. για τους στόχους 2020, προστασία του κλίματος, καταπολέμηση της κρίσης και βεβαίως υπάρχει σε όλα αυτά και η πολιτική της λιτότητας. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής, μπορείτε να μας εγγυηθείτε πώς θα υπάρξει ασφάλεια επενδύσεων για αυτούς τους ε, φορείς ε, δεδομένης δε και της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας. Και η μακροοικονομική αυτή αιρεσιμότητα, δηλαδή η διακοπή στην ανάγκη ε, της ε, χρηματοδότησης αυτής θα είναι μόνο η τελευταία δυνατή κίνηση. Σας ευχαριστώ. Απαντήστε. Σας ευχαριστώ. Ε, και εγώ από κάποια περιφέρεια κατάγομαι, από το ανατολικό κομμάτι της χώρας μου. Και ως, ε, και μάλιστα ήμουν μέλος ε, ενός οργανισμού που διέθετε περιφερειακά κονδύλια. Όσον αφορά λοιπόν την μακροερεσιμότητα των διαρθρωτικών ταμείων πρέπει να πω πως πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος. Ένα από τα διδάγματα της οικονομικής κρίσης είναι πως οι επενδύσεις αυτές πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε ένα υγιές μακροοικονομικό πλαίσιο για να μεγιστοποιηθεί ακριβώς ε, η χρήση των κονδυλίων. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να υπάρχει η ε, δυνατότητα να δημιουργούνται θέσει εργασία όταν χρησιμοποιούμε λεφτά των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Οι περιφέρειες λοιπόν παίζουν ένα σημαντικό ρόλο όταν μιλάμε για ε, νέα ανάπτυξη. Γιατί και οι επιτυχημένες εταιρείε ε, πάντα κάπου βρίσκονται. Και βεβαίως εξαρτώνται από το περιβάλλον τους παραδείγματο χάρη λεφτά τα οποία χρησιμοποιούνται για δεξιότητες κάπου σε μια περιφέρεια, για τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, για βασική έρευνα. Είναι χρήματα τα οποία εξοδεύονται σωστά και πρέπει να πάνε στα πανεπιστήμια, στους ερευνητές, στις επαγγελματικές σχολές μιας περιφέρειας. Γι' αυτό ακριβώς όπως είπα πολλές φορές έχουμε μια μακροοικονομική εμπιστοσύνη και τώρα πρέπει να στραφούμε προς την ανάπτυξη μαζί με τις περιφέρειες. Σας ευχαριστώ η κυρία Τιτσιάνα Μπέγκιν. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, εκτιμήσαμε τα όσα είπατε όσον αφορά την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Σχεδόν ξεχάσαμε σχεδόν ότι είστε ο ίδιος ε, Κατάινεν που είπατε όχι στην ε, Ελλάδα και απαιτήσατε εγγυήσεις. Ε, οι αξιολογήσεις θα πρέπει να ξεκινάνε από τα όσα έχουν γίνει ε, μέχρι στιγμής και δεν είναι θετικές. Για να είστε επίτροπος ε, πρέπει να γνωρίζετε την Ευρώπη, να είστε ευρωπαϊστής και να είστε ανεξάρτητος. Γνωρίζετε τις συνθήκες κύριε Κατάινεν, γιατί πριν ακόμα να δεσμευτείτε για τον προπολογισμό τα άρθρα της Ένωσης ε, ε, επιβεώνουν ότι προωθεί η Ένωση την ισότητα ανάμεσα στα κράτη, την ευημερία των πολιτών της. Ε, πώς αυτό το συνδυάζεται με τη λιτότητα και πώς εσείς δεσμεύεστε για την Ενωμένη Ευρώπη και για την αλληλεγγύη ακριβώς το αντίθετο από τα όσα ζητάτε. Ενώ εκατομμύρια Ευρωπαίοι χάνουν τη δουλειά τους, εσείς σε τέσσερις μήνες κερδίσατε σχεδόν 500.000 ευρώ μπορείτε να κάνετε αρκετά για την Ευρώπη. Σίγουρα κερδίζετε αρκετά. Διακόπτη ο Πρόεδρος. Είναι η σειρά του κυρίου Κατάινεν για να απαντήσει. Σας ευχαριστώ. Αν είμαι ο ίδιος Κατάινεν όπως ήμουνα, ρωτήσατε. Και αν θα προωθήσω τις βιώσιμες αξίες που χρειάζονται για να αυξηθεί το επίπεδο ε, ευημερία και ταυτόχρονα να αφημερινήσω για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Να σας διορθώσω για άλλη μια φορά. Μόνο ε, ήμουν υπεύθυνο. για το πέρασμα έξι πακέτων ε, δημοσιονομικής βοήθειας στη Φιλανδία. Μάλλον με μπερδεύετε με κάποιον από τους συναδέλφους σας εδώ που είναι από άλλα κόμματα και που ήταν κατά. Εγώ όμως παρουσίασα το πρώτο και δεύτερο ε, ελληνικό πακέτο στο Φιλανδικό Κοινοβούλιο και σας διαβεβαιώ πως δεν ήταν εύκολο. Κάποιοι φιλα... συνάδελφοι εδώ πολύ άγρια με, μου επιτέθηκαν. Και δεν ήταν εύκολο, αλλά κατά κάποιο τρόπο ήταν και εύκολο, διότι εγώ πίστευα πως ήταν ε, το σωστό αυτό που κάναμε από οικονομικής άποψης και από άποψη ελεγγύης. γι' αυτό είμαι ικανοποιημένος. Αν και κανείς δεν ήταν πολύ ε, ενθουσιασμένος με αυτά τα πακέτα οικονομικής βοήθειας. Τώρα, για την ευημερία και το κράτος πρόνοιας. Αυτό είναι στόχος για μας. Η οικονομία αγοράς είναι απλά ένα εργαλείο. Εκεί δεν υπάρχουν αξίες. Οι πολιτικοί πρέπει να δώσουν τις αξίες στην οικονομία της αγοράς. Και τώρα, όπως έχω ήδη πει, Πρέπει να εστιάσουμε στα συγκεκριμένα μέτρα που θα πείσουν τον ιδιωτικό τομέα να επενδύσει στην Ευρώπη και επίσης να επενδύσουμε στα συγκεκριμένα μέτρα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε τους δημόσιους, να χρησιμοποιήσουμε τους δημόσιους πόρους πιο αποτελεσματικά για να δημιουργήσουμε θέσεις. Η κυρία Πιετικάινεν είναι η επόμενη μιλήτρια. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα οικολογικά ε, όρια είναι συγκεκριμένα Ωραία, ε, το είναι πολύ συγκεκριμένα. Ε, αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε μια μισή φορά το πλανήτη μα, αλλά δεν μπορούμε να φτάσουμε στι τέσσερι φορέ, α πούμε. Το ίδιο ισχύει και με του προπολογισμού. Πρέπει να είναι αποτελεσματική όσον αφορά τις, τα έσοδα και τα έξοδα και θέλω να ακούσω πράγματα περισσότερα για τη στρατηγική σα πώ θα τα καταφέρετε και πώ θα λάβετε υπόψη το περιβάλλον και το ρόλο των ε, επιτρόπων αρμοδίων περί του κλίματος στον τομέα της οικονομίας. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πιετικάινεν. Αυτός ο τομέας είναι όντως ε, πολύ σημαντικός. Καταρχήν υπάρχουν κάποιες δημόσιες επενδύσεις, ε, δημόσιες μάλλον επιδοτήσεις με συγχωρείτε, που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά όσον αφορά τις βιώσιμες επενδύσεις. Εγώ έχω ασχοληθεί με αυτές τις μη υγιείς επιδοτήσεις σε διεθνές επίπεδο. Το θέμα είναι λοιπόν πώς μπορούν οι εθνικοί νομοθέτες να χρησιμοποιήσουν εργαλεία μέσα για να μπορέσουν να προωθήσουν την ανάπτυξη με οικολογικό τρόπο. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να δούμε μήπως κάποιες επιδοτήσεις από αυτές που δίνουμε δεν είναι βιώσιμες αποδοτικότητα των πόρων. Θα πρέπει να είναι τμήμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ε, να δημιουργήσουμε και πάλι τα εργαλεία για να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα και την αποδοτικότητα των πόρων. Επίσης θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε αν μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες καινοτόμες νέα καινοτόμα ε, δημοσιονομικά μέσα που να στηρίξουν την βιώσιμη ή την πράσινη ανάπτυξη. Η ε, Γενική Διεύθυνση Οικονομίας και Οικονομικών και η Διεύθυνση για το Περιβάλλον έχουν κάποιες ιδέες για το πώς θα συνδυαστούν τα δημοσιονομικά μέσα και τα συμφέροντα της πράσινης οικονομίας. Δεν είμαι πολύ εξοικειωμένος με τη θέση αυτή, αλλά θα τη μελετήσω περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γιούτα Στάινμπρουκ. Κύριε Κατάινεν, παρά τις με, μεταρρυθμίσεις, ίσως λόγω αυτών, η ανάπτυξη στην Ευρώπη και την Ευρωζώνη είναι χαμηλή. Εσείς είστε υποστηρικτής της πολιτικής λιτότητας που ε, είχε ως αποτέλεσμα απαράδεκτη ανεργία στην Ευρώπη. Το 2013 είχαμε 26 εκατομμύρια Ευρωπαίους ανέργους. Αυτοί δεν μπορούν. Δεν μπορούμε να τους πούμε ξεχάστε το παρελθόν. Οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται μέλλον ποια συγκεκριμένα μέτρα. Παρακαλώ να είστε συγκεκριμένος, είναι σημαντικό αυτό για την απόφαση που θα λάβουμε. Ε, ποια συγκεκριμένα πράγματα θα κάνετε για να επιτύχετε τους στόχους για την απασχόληση. Για να ε, καταπολεμηθεί η ανεργία και να βελτιωθεί και η ποιότητα της εργασίας. Κυρία Στάινρουκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Υπήρχαν αρκετές ερωτήσεις για το θέμα της ε, δημοσιονομικής πολιτικής και της εγγύησης των νέων και τις ε, ποιοτικέ θέσεις εργασίας των μέλλον. Ο μέλλον, ελπίζω, συνάδελφός μου, ο Πιέρη, είπε την προηγούμενη εβδομάδα πως πρέπει να μειωθεί το χρέος για να έχουμε ανάπτυξη. Και βεβαίως να έχουμε και μια ε, υγιή ε, δημοσιονομική πολιτική και κάθε ευρώ χρέους είναι ένα ευρώ λιγότερο για να επενδύσουμε στον τομέα της ε, υγείας ε, και στους Ευρωπαίους πολίτες. Πρέπει λοιπόν να βρούμε ένα πιο στοχευμένο τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα όπως η ανεργία των νέων. Η εγγύηση λοιπόν για την νεολαία είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα γιατί ήταν κάτι που δημιούργησε η κυβέρνησή μου και τώρα έχει αντιγραφεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και πράγματι νομίζω πως έχει φτάσει η στιγμή να δούμε το τι χρειάζεται ο κόσμος. Είναι πολύ στοχευμένο μέτρο. Δεν χρειάζονται όλοι το ίδιο φάρμακο. Αλλά αναλόγως με τις ανάγκες ε, των νέων θα δούμε αν θα πρέπει να εκπαιδευτούν ή κάπου αλλού να βρουν μια μαθητεία ή κάτι τέτοιο και σκοπεύουμε να το χρησιμοποιήσουμε πλήρως. Το θέμα είναι ότι χρειαζόμαστε θέσει εργασία ε, υψηλή ποιότητα, Γιατί έτσι ακριβώ θα έχουμε προστιθέμενη αξία. Σα ευχαριστώ. Ο κύριος Νότ Μαριάς. Εδώ κυρία Κατάινεν. Κύριε Κατάινεν, ήσασταν πρωθυπουργό της Φιλανδία και συμμετείχατε σε επίπεδο ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη λήψη των αποφάσεων για την επιβολή των καταστροφικών μνημονίων στην Ελλάδα η Ελλάδα μετά το μνημόνιο το Μάιο του 2010 και μέχρι σήμερα έχει λάβει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δάνεια ύψους 214 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και όμως έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Πώς το εξηγείτε αυτό. Πού πήγαν τα λεφτά κύριε Κατάινεν. Γιατί σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού της Ελληνικής Βουλής 2,5 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. 3,8 εκατομμύρια Έλληνες βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας λόγω υλικών στερήσεων και ανεργίας. Τα γνωρίζετε όλα αυτά. Αναλαμβάνετε την ευθύνη για την αποτυχία της πολιτικής σας και για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν νομίζετε ότι ήρθε η ώρα η Τρόικα να αποζημιώσει την Ελλάδα για την τεράστια οικονομική καταστροφή που προκάλεσε στην πατρίδα μου. Συγχωρείτε. Απα... Τελείωσε ο χρόνος σας, απαντήστε στην ερώτηση. Το θέμα δεν είναι αν μου αρέσει η ερώτησή σας, κατάλαβα τι λέτε, εντάξει. Ο ελληνικός λαός ε, έχει περάσει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση που έχουμε δει στην Ευρώπη και άλλο. Έχω φίλους που έχουν περάσει τα χειρότερα. Κάποιοι έχασαν τη δουλειά τους και μου κάνουν την ίδια ερώτηση. Πού πήγαν τα λεφτά. Ταυτόχρονα άλλοι λένε πως βοηθήσαμε την Ελλάδα με το να δανείσουμε διμερός. Και πάλι με ρωτάνε πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Ελπίζω τα θετικά μηνύματα που δεν φτάνουν ίσως στον απλό πολίτη, αλλά υπάρχουν το ότι δηλαδή η Ελλάδα έχει πρωτογενές πλεόνασμα και οι εξαγωγές προσπαθούν να ανακάμψουν και υπάρχει οικονομική ανάπτυξη ε, να συνεχιστούν και πρέπει να στηρίξουμε την Ελλάδα για να έχουμε ένα καλύτερο για να έχει ένα καλύτερο μέλλον. Γι' αυτό ακριβώς είναι σημαντικό αυτό το επενδυτικό πακέτο. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, ιδιωτικά και δημόσια, για να ενθαρρύνουμε τους επενδυτές να επενδύσουν και στην Ελλάδα. Η εμπιστοσύνη η οποία σιγά σιγά επανέρχεται στην Ελλάδα βοηθάει σε αυτή τη διαδικασία. Αλλιώ ο ιδιωτικό τομέα δεν θα μπορούσε να επενδύσει. Αλλά είμαι σίγουρο πω η κατάσταση θα βελτιωθεί πολύ τα επόμενα χρόνια και αντιλαμβάνομαι την, την δύσκολη κατάσταση στην Ελλάδα. Ε, Σας ευχαριστώ κυρία Κάλλας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε ένα χαρτοφυλάκιο που είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο με την ανάπτυξη, την απασχόληση και οι όροι είναι το βασικότερό μας μέλημα. Μας ενδιαφέρει λοιπόν η βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση. Πώς μπορούμε να επικεντρωθούμε στις ευφυείς επενδύσεις. Τι ακριβώς θα κάνετε για να είναι βιώσιμη η ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Ε, μία συνάδελφος λοιπόν και πρώην συνάδελφος και φίλη ε, Εσθονή που μίλησε φινλανδικά. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε για τις ευφυείς επενδύσεις όπως τις ε, κατονομάζουμε. Ο Κάρλος Μουέδας είναι ε, υπεύθυνος για τις ευφυείς επενδύσεις, δηλαδή τα ερευνητικά ταμεία. Πρόκειται για ε, μια μεγάλη πρόκληση για ολόκληρη την Επιτροπή, γι' αυτό χρειάζεται και ένα συντονιστικό ρόλο σε επίπεδο Επιτροπής, γι' αυτό δημιούργησε και αυτό το πρότυπο ο Ζαν Κλοντ Ιούνκερ αυτό έχει σημασία για την χρηματοδότηση της έρευνας. Έχουμε 80 δις για την έρευνα, υπάρχουν και άλλα ταμεία και τώρα θα πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτά τα ταμεία υπηρετούν την ανάπτυξη και τις ευφυείς επενδύσεις. Για παράδειγμα, οι ευφυείς μεταφορές για τους χρήστες ή επενδύσεις για το τομέα του περιβάλλοντος, ή ανανεώσιμες πηγές με βάση τα ανακυκλώσιμα υλικά ή και στον τομέα των ε, καυσίμων ή των οργανικών αποβλήτων θα πρέπει να ενισχύσουμε όλους αυτούς τους τομείς που άπτονται της έρευνας. Περιμένω λοιπόν πολλά από αυτή τη συνεργασία που θα ανακύψει και με τους άλλους ε, συναδέλφους, ιδιαίτερα τον Κάρλος Μουέδας και την Κρυσταλίνα Γεωργίεβα γιατί ασχολούνται με την κορονίδα του ζητήματος που αφορά δηλαδή την έρευνα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε υποψήφοι, Επίτροπε, συγκεκριμένα τι θα κάνετε για την πρωτοβουλία των κοινωνικών επιχειρήσεων και να εφαρμοστεί αυτή αποτελεσματικά. Γνωρίζετε πως ε, πρόκειται για έναν από τους λίγους κλάδους που επιδεικνύει άνοδο και είναι γύρω στο 10% της ευρωπαϊκής οικονομίας και βεβαίως αποδεδειγμένα έχει δυνατότητες ανάπτυξης για νέες θέσεις εργασίας, ειδικά για νέους. Τι θα κάνετε για να διευκολύνετε την ίδρυση νέων ε, τέτοιων κοινωνικών επιχειρήσεων και για την χρηματοδότησή τους και τι σκοπεύετε ε, να κάνετε ακριβώς ε, για να συντονίσετε τους τρεις συναρμόδιους επιτρόπους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ήταν εξαιρετική ερώτησή σας γιατί εξηγεί και ακριβώς το γιατί ο πρόεδρος Γιούνκερ θέλησε να δημιουργήσει αυτόν τον ε, ρόλο του συντονιστή των επιτρόπων. Τελειώσατε λέγοντας πως είναι διάφοροι επίτροποι συναρμόδιοι για αυτό το ζήτημα και για να αποφευχθεί η κλασική νοοτροπία ε, με τις παροπίδες πρέπει να συντονιστούμε πάρα πολύ καλά η ευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. και ενθαρρυντική. Και μ, αρέσουν, μ' αρέσει ένα συγκεκριμένο θέμα εκεί πέρα που είναι το ότι γίνεται αναφορά αναχώρα για τις πολυεθνικές. Είναι ένας ε, τρόπος καινοτόμος να μην έχουμε υπερβολική ρυθμισή, απλά να ορίζουμε πως οι μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες μπορούν να δημοσιεύουν ε, τις δραστηριότητές τους σε μια χώρα, το τι πήραν από αυτή τη χώρα και το τι πλήρωσαν. Αυτό είναι κατά την άποψή μου αντιπροσωπευτικό της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και νομίζω ε, έτσι ενισχύεται και η εμπιστοσύνη του κοινού ότι πληρώνονται ακριβώς οι φόροι αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Κυρία Κούμπουλα Νάτρη, θα κάνω δύο ερωτήσεις στα φιλανδικά για τον φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών και τους κοινωνικούς δείκτες. Κύριε Κατάινιν, και εγώ είμαι υπερήφανος για την ε, φιλανδική εγγύηση των ε, νέων, αλλά δεν είμαι υπερήφανη για αυτά τα οποία έγιναν με τον φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Είναι η τρίτη φορά που σας έγινε αυτή η ερώτηση. Μπορείτε λοιπόν να απαντήσετε. Κυρία Τάισεν μίλησε και είπε πως θα ληφθούν υπόψη και οι κοινωνικοί δείκτες όταν μιλάμε για μακροοικονομικές ανισορροπίες. Γνωρίζετε αυτά τα ζητήματα από τη Φιλανδία. Οι προτάσεις του προπολογισμού ποτέ δεν γίνονται χωρίς να ληφθεί υπόψη ε, ε, ο αντίκτυπος στην απασχόληση και αλλού. Μπορείτε να μας δώσετε και, την ίδια, και εσείς την ίδια υπόσχεση όπως η κυρία Τάισεν. Σας ευχαριστώ για τον φόρο αυτόν. Η Κομισιόν έκανε μία πρόταση στις χώρες που θέλουν να συνεργαστούν σε αυτό. Και ο ρόλος της είναι αυτή τη στιγμή να διασφαλίσει πως δεν θα εμποδίσει τις χώρες οι οποίες θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Αυτό τώρα θα το αποφασίσουν τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν είναι σε θέση να βοηθήσει. Η Φιλανδία τώρα δεν ήθελε για τους ίδιους λόγους που δεν ήθελε και η Σουηδία. Φαντάζομαι πως δεν θέλουμε να το συζητήσουμε περισσότερο, επί η Σουηδία όχι, είπαμε και εμείς όχι. και μάλιστα εισήχθη ένα τέλος σταθερότητας στις ε, τράπεζες που μοιάζει πάρα πολύ με το τέλος που επιβλήθηκε στην ε, Σουηδία και αυτό οδήγησε στο ότι κάποιες τράπεζες ε, μετέφεραν στοιχεία τους από τη Φιλανδία στην Σουηδία. Δεν θέλω να το επαναλάβω αυτό, δεν θα ήθελα εγώ να κάνω κάτι για να χάσει τη δουλειά του κάποιος υπάλληλος τράπεζας. Εάν όλοι το κάνουν όλες οι χώρες, τότε ναι, να το δεχτούμε. Μετά, για τους δείκτες της ε, απασχόλησης. Αυτό πρέπει να το δούμε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αλλά από την άλλη πρέπει να δούμε προσεκτικά το εάν η διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών είναι το σωστό μέρος για να δούμε τους κοινωνικούς δείκτες, γιατί χρειαζόμαστε δείκτες που θα μας βοηθήσουν για τις μελλοντικέ κρίσεις σε 5 ή 10 χρόνια. Εάν αυξηθεί η ε, ανεργία, θα το δούμε, αλλά τα προβλήματα αυτά υπάρχουν τώρα. Δεν είναι κάτι το οποίο θέλουμε στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Αρβαζά. Κύριε Χέρνα Βίρκουνεν, κύριε Κατάινεν, ο νέας σας ε, τομέας ε, οι επενδύσεις και η απασχόληση είναι κάτι που σας είναι οικείο. Στη Φιλανδία, στη πάντα ε, ταχθήκατε υπέρ των επενδύσεων στην έρευνα, την επιστήμη και την εκπαίδευση και μιλήσατε για την πράσινη ανάπτυξη, μιλήσατε και για το πράσινο αυτοκίνητο και τις πράσινες μεταφορές γενικότερα οικολογικές μεταφορές. Τώρα θα πρέπει να προωθήσετε την οικονομική, την ε, οικονομική ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζετε, πού θα πρέπει να επιτύχει η Ευρώπη για να δημιουργήσει ε, ανάπτυξη. Απάντηση. Το πιο σημαντικό είναι να αρχίσουμε από την σταθερότητα. Θα πρέπει να μην υπάρχουν αμφιβολίες από τα κράτη-μέλη ως προς τις ε, δυνατότητες ανταπόκρισης. Η Ευρώπη θα πρέπει να φανεί δυνατή στην Ευρώπη και να παράξει εμπιστοσύνη, να δημιουργήσει εμπιστοσύνη. Επίσης θα πρέπει να έχουμε τα δημόσια μέσα, τους δημόσιους πόρους για ένα νέο κύμα επενδύσεων. Και φυσικά να διοχετεύσουμε και τις ε, ιδιωτικές επενδύσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να επενδύσουμε στην έρευνα και την ανάπτυξη. Το ίδιο αφορά και τα πανεπιστήμια. Ακόμα και αν οι επιπτώσεις στην απασχόληση δεν φαίνονται άμεσα. Νομίζω όμως ότι θα υπάρξει αναγέννηση στην Ευρώπη από την έρευνα και την ανάπτυξη. Ως προς την ενέργεια και τις μεταφορές δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ενεργειακή προμήθεια και ασφάλεια είναι ύψης της σημασίας για τα νοικοκυριά αλλά και για τις βιομηχανίες και πρόκειται για έναν τομέα που δεν υπάρχει ακόμα εσωτερική αγορά στην ψηφιακή αγορά δεν υπάρχει ακόμα ε, ενποιημένη εσωτερική αγορά. Ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει στις ίπα, Γιατί μιλάμε για 300 ε, εκατομμύρια πιθανούς χρήστες ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 28 διαφορετικά συστήματα. Υπάρχει κατακαιρματισμός της αγοράς. Θα πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες για να δημιουργήσουμε μία εσωτερική και ενεργειακή ε, αγορά, ιδιαίτερα ψηφιακή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κατάινεν. Όπως γνωρίζετε, μία ε, βασική δέσμευση του Πρόεδρου Γιούνκερ είναι τα 300 δις, ε, το επενδυτικό αυτό πακέτο για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση και οι περισσότερες ερωτήσεις κατευθύνθηκαν σε αυτό το πακέτο. Πώς μπορείτε να μας εγγυηθείτε ότι θα υπάρξουν νέοι πόροι από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με διάφορα μέσα, διότι υπάρχει υποψία ότι θα γίνει μια επαναδιανομή των χρημάτων που ήδη διατίθενται. Και πώς βλέπετε το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής αυτού του προγράμματος. Ποια είναι τα συγκεκριμένα μέσα και πού θέλετε να προβείτε στην επαναβιομηχάνηση της Ευρώπης, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον της. Ευχαριστώ πολύ. Απάντησε. Μιλήσατε για το χρονοδιάγραμμα και για το πώς θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε πραγματικές επενδύσεις, όχι επενδύσεις επί χάρτου και τι μπορούμε ε, να κάνουμε για την ε, εκ νέου εκβιομηχάνηση της Ευρώπης. Ως προς το χρονοδιάγραμμα ή τον χρονισμό μάλλον εφαρμογής των μέτρων. Αυτό αφορά ε, συγκεκριμένους τομείς, δηλαδή στην Ενεργειακή Ένωση ή την ψηφιακή αγορά. Εάν υπάρχουν επενδύσεις στα ευρυζωνικά συστήματα, για παράδειγμα, τότε θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, αλλά η τελική ε, έκβαση, το τελικό αποτέλεσμα μάλλον, δεν αφορά τα ευρυζωνικά συστήματα, αλλά καλύτερο περιβάλλον για την ανάπτυξη των βιομηχανιών. Και αυτό το πλαίσιο είναι λίγο διαφορετικό, διότι τίνει σε ε, υπάρχουν τα χρηματοοικονομικά μέσα δηλαδή η ΕΤΕ, ε, έχει μεγαλύτερη δυνατότητα δανειοδότησης πλέον. Πολλοί λένε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πιο αποδοτικά ο κοινοτικό προπολογισμό, γιατί ανακυκλώνουμε το ε, χρήμα. Αν δεν κάνουμε τίποτα, τότε ξέρουμε το αποτέλεσμα. Αν αλλάξουμε όμως προτεραιότητες, μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα. Άρα θα υπάρχει νέο, φρέσκο ε, δημόσιο χρήμα και από αυτό το τομέα. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να ιεραρχήσουν τις επενδύσεις όχι μόνο για την αρχική όθηση, αλλά και για τη δική τους οικονομία. Οι περισσότερες ε, ε, ερωτήσεις έχουν υποβληθεί από τις τρεις επιτροπές. Τώρα η Επιτροπή Μεταφορών θα υποβάλει ερωτήσεις. Μάρκος Πίπερ. Ναι, κύριε Κατά Κατάνιν, καμιά φορά έχει κανείς την εντύπωση πως θα δώσουμε περισσότερα λεφτά από την Ευρώπη και όλα θα πάνε καλά στη διαρθρωτική πολιτική, στη γεωργία, παντού. Μπορεί κανείς να διαφωνεί, αλλά μπορεί να πει κανείς πως όσο δεν μπορούν να αντλήσουν τα κράτη-μέλη τα κονδύλια παρκώς, δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν σωστά και μια φορά άλλα τέτοια υπάρχει, ε, υπάρχουν ακόμα κάποια διαθέσιμα τα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε σε συνδυασμό με ιδιωτικά κεφάλαιο, Ένα ερώτημα. Τι μπορείτε να κάνετε για να δημιουργήσετε ως συντονιστής συνθήκες ανάπτυξης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ως αντιπρόεδρος που συντονίζετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πρώτο σας ερώτημα ήταν πώς να αποφύγουμε την κακή χρήση των δημοσίων πόρων και πράγματι χρειάζεται μια ανάλυση κόστους ωφέλους πριν ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο. Τα λεφτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς και διάφορους τρόπους αποτελεσματικούς ή όχι τόσο. Η πρόκληση είναι πόσο μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να μπορέσουν να πάρουν και αυτές ε, δημόσια έργα. Και μία απάντηση είναι ένα πιο διαφανές σύστημα δημοσίων προμηθειών. Και έτσι θα μειωθεί και η διαφορά. Εύκολα μπορούμε να αντιληφθούμε πως ε, υπάρχουν πολλές καινοτόμες μικρομισές επιχειρήσεις που είναι διατεθειμένες ε, να πάνε και να κάνουν μια προσφορά για ένα δημόσιο έργο εάν ξέρουν πως θα είναι δίκαιος ο ανταγωνισμός. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε ήδη συζητήσει με τον Επίτροπο τον Αρμόδιο για την Ενιαία Αγορά. θα είναι αυτό ένα σημείο στο οποίο θα εστιάσουμε. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Εύα Καϊλή. Πέρα από τους ευσεβείς πόθους μπορείτε να μας δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις. Είστε ικανοποιημένος για το ότι η Ελλάδα επέστρεψε στις αγορές πέρα από το 27% της ανεργίας, ε, την ύφεση και τη μείωση των μισθών που δεν αποκατέστησε την ανταγωνιστικότητα στι νότιε χώρε. Πρέπει να κόψουμε κι άλλο. Η αγαπημένη σας ε, λιτότητα είναι ο μόνος τρόπος για ανάπτυξη από τη λέτε. Είναι ηθική. Μήπω ε, ε, θα σα ικανοποιούσαν λιγότερες ε, θυσίες από τους φτωχού, Διαφωνείτε με τον κύριο Γιούνκερ ο οποίος είπε λιγότερες ε, προδιαγραφές. Και επιπλέον, εάν όμως κοβησεί διαλέξει μια διαφορετική πολιτική από εσάς, θα προσπαθήσετε να τον σταματήσετε ως συντονιστής ή θα προσπαθήσετε ε, να δεχτείτε αυτά τα οποία λένε οι υπόλοιποι επιτροποί χωρίς να μας πατρονάρετε εμάς τους νότιους. Μπορείτε σας παρακαλώ να είστε πιο αξιόπιστος και πιο συγκεκριμένος. Ευχαριστώ. Πολλές μια μεγάλη που δεν έχει απαντηθεί. για το εάν θα ακολουθήσω τη γραμμή Μοσκοβησία αν έχουμε διαφορετικές απόψεις και το εάν είπα ότι η λιτότητα είναι ο μόνος τρόπος για ανάπτυξη. Πρώτα απ' όλα εγώ δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο γιατί δεν το πιστεύω. Δεν ξέρω γιατί ε, είπε κάποιος κάτι τέτοιο. Εγώ ξέρω πως δεν έχω πει ποτέ κάτι τέτοιο. Είμαι 100% σίγουρος. Αυτό το οποίο πιστεύω είναι πως τα δημόσια οικονομικά πρέπει να είναι υγιή ακριβώς για να υπερασπίσουμε και το κράτος πρόνοιας. Και όπως είπε και ο Γιούνκερ, δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε κράτος πρόνοιας με όλο και μεγαλύτερο χρέος. Και συμφωνώ πλήρως με αυτό το οποίο είπε ο Πιέρο, ότι κάθε ευρώ που ξοδεύεται για την εξυπηρέτηση του χρέους αφαιρείται από τον κόσμο. Οπότε χρειάζεται και καλύτερη, πιο αξιόπιστη πορεία, αλλά ταυτόχρονα χρειαζόμαστε πιο συγκεκριμένες επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Εγώ θα επικεντρωθώ τώρα στα ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη, όχι τόσο την ε, δημοσιονομική πολιτική. Δεν ε, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ε, ένας άλλος αντιπρόεδρος, ο Βαλτές, θα συντονίζεται με τον Πιέρ. Ο Βάλτης Ντομπρόφσκης θα ασχοληθεί με αυτό το ε, θέμα. Εγώ θα συντονιστώ με τον Πιέρ για τη δημιουργία θέσεων ε, εργασίας και νομίζω πως ε, είναι και καλύτερο το δικό μου χαρτοφυλάκιο. Président, Monsieur le Commissaire désigné votre. Ευχαριστώ πολύ γιατί μας ε, μιλήσατε για την ε, εμπειρία σας ως ε, Πρωθυπουργού της Φινλανδίας και σε αυτά τα πλαίσια προσπαθήσατε να καταπολεμήσετε την ανεργία των νέων. Αυτό σας έδωσε και μία σαφή νομιμότητα. Έχουμε τα μέσα πώς μπορείτε ως ε, ε, αρμόδιος να τετραγωνίσετε τον κύκλο, ε, δηλαδή να ασχοληθείτε με τις νέες θέσεις εργασίας και από την άλλη πλευρά να ανταποκριθείτε στην ανεργία των νέων, ιδιαίτερα αυτούς που δεν έχουν ε, ιδιαίτερα προσόντα ή δεξιότητες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, πρόκειται για ένα πολύ συγκεκριμένο ένα πολύ συγκεκριμένο μέσον, γιατί στην Αυστρία υπάρχει ένα ειδικό ε, θέμα ε, μαθητείας, πρόγραμμα μαθητείας και αν ήμουν πρωθυπουργό, ακόμα πρωθυπουργό, θα ε, ήθελα να μιμηθώ αυτό το αυστριακό πρότυπο για τη μαθητεία στους νέους. Εμείς ε, δεν έχουμε μιλήσει για το ρόλο των νέων στην αγορά εργασίας ε, τόσο πολύ. Νομίζω θα πρέπει να συμμετάσχουν και οι γυναίκες περισσότερο στην αγορά εργασίας. Είναι ένα θέμα ισότητας και οικονομικής ανάπτυξης. Ένα άλλο θέμα είναι ότι θα πρέπει να προσδώσουμε μεγαλύτερη σημασία ε, στους ανάπηρους, ε, δηλαδή στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, γιατί δεν πρόκειται μόνο για απόκτηση χρημάτων, αλλά για το πώς μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί, να βοηθήσουμε τους πλέον ευάλωτους και αδύνατους και τα ίδια δικαιώματα αφορούν τους, ε, τα άτομα με ειδικέ ανάγκες. Ε, όταν ήμουν ε, Πρωθυπουργό, συντάξαμε ένα πρόγραμμα 18 εκατομμυρίων ευρώ έτσι ώστε οι εργοδότες να προσλαμβάνουν αμαία. Το πρόγραμμα λειτουργήσε πολύ καλά και εκτιμήθηκε δεόντως. Άρα υπάρχουν ε, ε, ζητήματα για το τι μπορούμε να μάθουμε οι μεν από τους δε. Και νομίζω ότι θα πρέπει και η Επιτροπή να ε, ασχοληθεί και να αντιγράψει τις καλύτερες πρακτικές. Από την Ρέγκη, Κωνσταντς Ρέιου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κατάινεν, θα είστε επίσης υπεύθυνος για τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής και Πολιτικής Έρευνας. Ποια συγκεκριμένα μέτρα βλέπετε για να εξασφαλίσουμε τις ε, μέγιστες συνέργειες σε αυτόν τον τομέα και τι θα κάνετε για να στηρίξετε τις περιφέρειες για να εξειδικευτούν και θα επανέλθω σε αυτά τα 300 δισεκατομμύρια το επενδυτικό πρόγραμμα λέτε πως έχετε πρόθεση να διαθέσετε κονδύλια της διαρθρωτικής πολιτικής τα οποία έχουν ήδη διατεθεί και να πάνε αυτά στο πρόγραμμα επενδύσεων της Κομισιόν ενώ έχουν ήδη δεσμευτεί αλλού. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει ακόμα η νέα επιτροπή, δεν έχει συσταθεί. Όμως έχουμε συζητήσει με την Κρυσταλίνα για τη χρηματοδότηση της έρευνας μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ε, προϋπολογισμού, το πρόγραμμα του Horizon. Υπάρχουν αρκετά χρήματα για την έρευνα αλλά ε, υπάρχουν και 15 διαφορετικές γραμμές του προϋπολογισμού για να υποστηρίξουμε την έρευνα στις ΜΜΕ ιδιαίτερα. Επίσης χρησιμοποιούμε τα χρήματα από τα διαρθρωτικά ταμεία για τις έρευνες. Η κρυσταλλίνα είναι πλέον αρμόδια επί του θέματος, αλλά πιστεύω αυτά που μου είπε, ότι θα πρέπει δηλαδή όλα αυτά να τα δούμε με μεγάλη προσοχή ως προς τη χρήση των διαρθρωτικών ε, ταμείων για να δούμε πώς ε, μπορούν να συγχωνευτούν γραμμές του προϋπολογισμού για να ε, έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Και η ΕΤΕ θα πρέπει να συμμετάσχει ή άλλα χρηματοοικονομικά μέσα. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και με τα διαρθρωτικά ταμεία και με τον ορίζοντα και ίσως και ιδιωτικούς πόρους. Είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Βέρνερ Λάγκεν. Ευχαριστώ κύριε Κατάινεν. Θα ήθελα να συμφωνήσω με την Λίζα Φερέρα. Πρέπει να σας μετράμε με βάση τις πράξεις σας. Και εδώ πέρα πραγματικά η Φιλανδία είναι μια σύγχρονη χώρα με χαμηλό χρέος, βιομηχανία, ε, έχει επιτύχει τις ίσες αμοιβέ ανδρών και γυναικών, μα έπρεπε να είναι ιδεώδης χώρα των αριστερών. Και παρόλα αυτά σας ζητάνε να υποβάλλετε συνταγές ε, για το πώς θα πετύχετε πράγματα μαγικά. Κοιτάξτε, μας λένε οι αγορές ξεκάθαρα πως ε, το όριο έχει φτάσει σε ένα χρέος, έχει σε ένα, το χρέος μας έχει φτάσει σε ένα όριο, στο μη περαιτέρω. Και βεβαίως αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να κινητοποιήσουμε το ε, ιδιωτικό κεφάλαιο για να πάει σε επενδύσει αντί να κρύβεται στο, σε hedge funds στο Λουξεμβούργο, Συγκαπούρη και αλλού. Τι σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Λέτε πως το σημαντικότερο είναι να βρούμε περισσότερα χρήματα για πραγματικές επενδύσεις και να μην μένουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Άρα δεν είναι μόνο θέμα ρευστότητας. Διότι δεν μας λείπουν ε, χρήματα. Κοιτάξτε, πρέπει να πούμε ξεκάθαρα πως μας λείπει και η ζήτηση και η προσφορά. Τώρα το ότι ήμουν ε, πρωθυπουργό σε μια κυβέρνηση με κόμματα και γκουε και φιλελευθέρων και ΕΛΚ, νομίζω πω με κάνει κάποια πράγματα να ξέρω για τη συνεργασία. Γνωρίζω παραδείγματο χάρη το ότι εάν αρχίσει κανείς να προκαλεί τις εταιρείε του με τι οποίε πρέπει να συνεργάζεται, δεν βοηθάει. Το είχαμε ξεκινήσει αλλά μετά σταματήσαμε γιατί κάθε φορά που ξεκινούσαμε καυγάδε χρειάζονταν ώρες μετά για να λυθούν τα προβλήματα. Θα ήθελα ακριβώ και εγώ να βοηθήσω για να υπάρχει μια συνεννόηση έτσι ώστε ο κ. Λάγκεν, η κυρία Φερέιρα και εγώ να βρούμε κάποια πράγματα που μα ενώνουν. Υπάρχουν αρκετά προφανώ που μα χωρίζουν. Αλλά Ε, μπορώ να σου πω δέκα πράγματα που μας ενώνουν και να εστιάσουμε σε αυτά. Ας επικεντρωθούμε λοιπόν στα ζητήματα που μπορούν να μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο. Σας ευχαριστώ. Γιένς Νίλσον από την Επιτροπή Μεταφορών. Εδώ είμαι, πίσω πίσω. Επανέρχομαι σε αυτό που ήδη έχει αναφερθεί. Ήδη άλλοι επίτροποι το απάντησαν για το κοινωνικό ντάμπινγκ, ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών. Ήταν μια βασική αίτηση για τον αθέμητο ανταγωνισμό και το κοινωνικό ντάμπι που βλέπουμε στις μεταφορές σε παγκόσμιο επίπεδο και συγκεκριμένα οι οδικές μεταφορές. Αντιπρόεδρος ε, με την ευθύνη για τον συντονισμό της πολιτικής μεταφορών. Αυτό προβλέπεται για σας, αλλά δεν άκουσα πραγματικά κάτι συγκεκριμένο, γι' αυτό πιστεύω ότι είναι απαραίτητη η απάντηση. Τι θα κάνετε για να βάλετε στην προτεραιότητα την καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ στον τομέα των μεταφορών. Ευχαριστώ. Thank you Σα Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Έχετε μεγαλύτερη εμπειρία στον τομέα αυτό από ότι εγώ. Η αρχή θα πρέπει να είναι ότι αν ακόμα και όταν κάνουμε πανευρωπαϊκές επενδύσεις για τις μεταφορές, η υποχρέωσή μας είναι να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία για ολόκληρη την Ευρώπη, να συνδέσουμε δηλαδή τον κόσμο και τις αγορές καλύτερα από ό,τι πριν. Ενώ η προϋπόθεση για τη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων θα πρέπει να είναι ότι οι επενδύσεις πληρούν όλα τα κριτήρια που χρειάζονται στην κοινωνική οικονομία της αγοράς. Και η κοινωνική, το κοινωνικό dumping δεν μπορεί, δεν έχει χώρο εδώ. Ε, αν υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις σε τέτοιου είδους συμπεριφοράς, ευχαρίστως θα ήθελα να ακούσω περισσότερα, διότι πρέπει να αναπτύξουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να αναγνωρίζουμε καλύτερα τέτοια στοιχεία και να αντιμετωπίσουμε. Εάν υπάρχουν ε, στοιχεία γκρίζας οικονομίας, η παραοικονομίας, να μπορούμε εύκολα να τα ε, εξοπελίσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω κι άλλα στοιχεία. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση. Μπούρχαρτ Μπάιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Κατάινεν. Θα ήθελα να θέσω τρία σύντομα ερωτήματα. Πρώτον για το ευρωπαϊκό εξάμεινο, ειδικά στον αφορά τις συστάσεις αναχώρα. Ως αντιπρόεδρος είστε αρμόδιος για την ανταγωνιστικότητα. Πώς θα διασφαλίσετε πως ε, θα παίξει σημαντικό ρόλο η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στις συστάσεις αυτές. Δεύτερη ερώτηση. Χαιρετίζουμε αυτό το οποίο είπατε πως πρέπει να υπάρξει ενίσχυση των επενδύσεων αλλά βεβαίως οι επενδύσεις έχουν και κινδύνους πως θα τους αντιμετωπίσετε αυτούς και τέλος είπατε πολλές φορές πως θέλετε να συνεργαστείτε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πως θα εγγυηθείτε τη συναπόφαση του Ευρωπαϊκού πακέτου στο, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πακέτο των επενδύσεων Ευχαριστώ Thank σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν το πρώτο σας ερώτημα ήταν οι συστάσεις προς τα κράτη-μέλη. Από ό,τι θυμάμαι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέλησε ε, με βάση την εφαρμογή του 18% των CSA. Υπάρχουν πιο ε, αισιόδοξα ή πιο απεσιόδοξα στοιχεία αλλά εν πάση περιπτώσει ε, θα χρειαστώ τη βοήθειά σας ε, για την έμπρακτη εφαρμογή. Γιατί εσείς μπορείτε να επηρεάσετε τη χώρα σας. Εγώ θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να ενισχύσω το θέμα αυτό των συστάσεων, διότι πρόκειται για ένα μέσον που αφορά ε, καθαρά νομοθετικό έργο τα CSR εντάσσονται στο ευρωπαϊκό εξάμεινο και οπωσδήποτε ε, αποκτούν μεγαλύτερη σημασία αυτές οι συστάσεις αναχώρα. Εάν εμπλέκεται ο ιδιωτικός τομέας, τότε ε, υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος, ο όμως, τον οποίο όμως θα πρέπει να επομιστεί ο δημόσιος τομέας. αλλά αν υπάρχει κοινοπραξία τότε θα πρέπει να υπάρχει επιμερισμός κινδύνου. Γι' αυτό θα πρέπει να μειωθεί το επίπεδο κινδύνου, ιδιαίτερα στις υποδομές δηλαδή. Το ιδιωτικό χρήμα, οι ιδιωτικές πηγές δεν θέλουν να αναλάβουν τόσο υψηλό κίνδυνο. Γι' αυτό χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε ε, δημόσιους πόρους για την εξισορρόπηση. Επίσης θα πρέπει να βελτιστοποιήσουμε τον, ε, την συμμετοχή των κρατών. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους από ΙΤΡΕ, ΕΚΟΝ και από την, στις μεταφορές και την ΡΕΓΙ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλες τις επιτροπές Εμπλήτρε και Έκον και τώρα ο, υποψήφιος μπορεί να ε, προβεί σε μια καταληκτική ε, δήλωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Είναι η πρώτη φορά που είχα την ευκαιρία να ξανασκεφτώ το ζήτημα του πακέτου των επενδύσεων, της ανάπτυξης και της απασχόλησης. αν ε, εγκριθεί ο διορισμός μου, θα ήθελα να ξανασυζητήσουμε τις προτεραιότητες της κάθε επιτροπής, του καθένα, ποιες θα είναι οι προτεραιότητες του πακέτου επενδύσεων και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα ο κοινοτικός προϋπολογισμός και ποια χρηματοοικονομικά μέσα θα θέλατε και μέτρα θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε περισσότερο. Επίσης, εάν με εγκρίνετε, θα ήθελα τη βοήθειά σας για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, ε, ιδιαίτερα σε θέματα που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά. Ε, πολλά κράτη αντιτάχθηκαν, αλλά τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα για πιο φιλόδοξες ε, προσπάθειες για να δημιουργήσουμε μία πραγματικά ενιαία αγορά, να βοηθήσουμε τις ε, ΜΜΕ να προωθήσουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους. Όπως σας είπα και πριν, θα ήθελα να καταβάλω προσπάθειες για πραγματικές επενδύσεις και πραγματική συνεργασία ε, παρόλο που δεν είμαι πολιτικός ε, πλέον, είμαι δημόσιος υπάλληλος. Ξέρω ότι πολλές φορές υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ ζητημάτων και αξιών. Αλλά πολλές φορές οι πολίτες, ε, στους πολίτες δεν γινόμαστε αρεστοί όταν δίνουμε μάχες ως πολιτικοί. Γιατί να μην επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα θέματα που μας βρίσκουν σύμφωνους. Δυστυχώς δεν έχει επανέλθει η εμπιστοσύνη στους πολίτες, στον κοινό μέσο άνθρωπο. Δεν θα ήταν σκόπιμο λοιπόν να δημιουργήσουμε τις συνθήκες, τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε να βρούμε τα ζητήματα που μπορούν να μας βρουν σύμφωνους και όπου δεν υπάρχει διαφωνία και να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία και αυτό το πνεύμα συνεργασίας για να προωθήσουμε τις επενδύσεις, ε, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω λοιπόν για αυτή την εξαιρετική ανταλλαγή απόψεων. Σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο εβδομάδας και ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Μιλώ γρήγορα πολλές φορές, γι' αυτό σας ευχαριστώ όλους και το Προεδρείο καθώς και τη Γραμματεία για αυτή την ευκαιρία που μου δώσατε να εκφράσω τις απόψεις μου. Ευχαριστούμε κύριε υποψήφιε επίτροπε. Θα ήθελα ο κύριος Γκουαλτιέρη να λάβει το λόγο για ορισμένα τελικά σχόλια. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον υποψήφιο επίτροπο Κατάινεν για την ενδιαφέρουσα ακρόαση τα μέλη της ΕΚΟΝ καθώς και την ΙΤΡΕ. Ε, Θα ήθελα τα μέλη της ε, ΕΚΟΝ να μεταβούν στην ακρόαση του κυρίου Χιλ. Δίνω το λόγο στη Μαρίτα Ολσκοπ. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τις ερωτήσεις σας και τον κύριο Κατάινεν ιδιαίτερα για τις απαντήσεις του. Περάσατε δύσκολες ώρες, αλλά νομίζω ότι έτσι έχει η διαδικασία των ακροάσεων και φτάνουμε και στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά αυτόν τον τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την ακρόαση αυτή και δεν είναι και η τελευταία να το τονίσω αυτό. Ευχαριστώ τους συμπροέδρους και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους τα μέλη του ε, Ευρωκοινοβουλίου. Τώρα ορισμένε ε, πληροφορίες στις 2.30 έχουμε την ακρόαση του κυρίου Τίμερμανς, υποψηφίου αντιπροέδρου. Επίσης διάσκεψη των ε, προέδρων που είναι ανοιχτή σε όλους. Θα πρέπει να είμαστε παρόντες. Επίσης, στη μια μισή οι συντονιστές της ΙΤΡΕ Econ Employment, στις 6, στις 6 αυτό. Και στις 7 συνεδρίαση με την ΕΜΒΗ. Ευχαριστώ και την κοινή γνώμη που μας παρακολουθεί και βρίσκεται κοντά μας. Σας ευχαριστώ όλους.